Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ θα μιλήσω γαλλικά. Βάλτε τα ακουστικά σας τώρα. Καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω και να καλωσορίσω την κυρία υποψήφια επίτροπο στην ακρόση αυτή που είναι η πρώτη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θα ακούσουμε επίσης δύο επιτρόπους και έναν εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή είναι η πιο πολυπληθής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή τη θητεία Νομίζω ότι κυρία υποψήφια επίτροπε αυτό είναι σαφές μήνυμα για τη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας αλλά που θα σα απασχολήσουν φυσικά και εσάς διότι στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της ε, κυρίας Φόντερ Λάιεν υπάρχουν τα θέματα φυσικά υγεία, το σχέδιο δράση κατά του καρκίνου αλλά και τα θέματα ασφάλεια τροφίμων της καταπολέμησης της μόλυνσης και της στρατηγικής από το χωράφι στο πιάτο. Πολλά θέματα λοιπόν που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Επιτρέψτε μου κυρία υποψήφια επίτροπε μία παρατήρηση πριν σας δώσω το λόγο και, και αφού φυσικά εξηγήσω τη διαδικασία. Τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος με τα οποία εδώ και μέρες συζητώ από τότε που λάβαμε τις γραπτές απαντήσεις σας συμμερίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό μία άποψη. Την άποψη ότι για το τμήμα της υγείας των απαντήσεών σας υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λοιπόν έχει να κάνει και με την προσωπική σας ε, σταδιοδρομία. Αντίθετα, τίθενται ερωτήματα για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων ιδιαίτερως. Εκρίθησαν βέβαια, θα επανέλθουμε, εκρίθησαν πολύ πιο γενικόλογες. Σας το λέω λοιπόν ήδη, γιατί ήδη είχαμε προηγουμένως ε, μία ακρόαση με τον ε, υποψήφιο για την Γεωργία που θεωρήθηκε ιδιαίτερα γενικόλογο. Αναμένουμε λοιπόν από εσά συγκεκριμένες απαντήσεις, τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα σας τεθούν από τα μέλη της Επιτροπής μας. Τώρα, πώ θα λάβει η χώρα η συζήτηση. Οι συντονιστές έκαναν μια μικρή προσαρμογή στη διαδικασία, δηλαδή ο καθένας μας θα έχει 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα για να κάνει ερωτήσεις. Κατόπιν, η κυρία υποψήφια επίτροπος θα έχει 2 λεπτά για να απαντήσει. Κατόπιν, 45 δευτερόλεπτα, μέγιστο, για μια συμπληρωματική ερώτηση. Και επιμένω ότι μας έχει ζητηθεί οι συμπληρωματικές ερωτήσεις να είναι πραγματικά συμπληρωματικές ερωτήσεις, διευκρινιστικές. Δηλαδή να είναι συνέχεια της προηγούμενης, της πρώτης ερώτησης για να διευκρινιστεί η απάντηση. Όχι για να ξεκινήσει μια συζήτηση για ένα άλλο θέμα γιατί η κυρία υποψήφια επίτροπος θα έχει μόνο ένα λεπτό για να απαντήσει. Θα είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να περάσουμε με σαφή και κατανοητό τρόπο σε ένα άλλο θέμα. Παρακαλώ να σεβαστείτε όλοι ε, το πνεύμα αυτής της διαδικαστικής προσαρμογής. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία υποψήφια επίτροπο για 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΕΜΒΗ και Άγκρη, κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα ενώπιαν των ερετών δημοκρατικά εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αναζητήσω την επιβεβαίωσή σας ως Επίτροπος Αρμόδιος για την Υγεία. Επιτρέψτε μου όμως να πω δύο λόγια στην γλώσσα μου, στα ελληνικά. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα σαν υποψήφια Επίτροπος Υγείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα θέματα υγείας αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει για μένα την πηξίδα που θα με καθοδηγεί κατά τη διάρκεια της θητείας μου σαν Επίτροπος, εάν επιβεβαιωθώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Dear friends and colleagues. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν να υπάρχει πρόσβαση στην υγεία, ασφαλή τρόφιμα και προστασία κατά των επιδεμιών και των νόσων για να νιώσουν ήρεμοι. Το αξίζουν αυτό. Έχουμε κάποια από τα υψηλότερα πρότυπα σε θέματα φυτοϊγείας και υγείας των ζώων και τα καλύτερα συστήματα υγείας, τα οποία είναι προσιτά σε όλους και προσβάσιμα σε όλους, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις προσδοκίες, για να μην έχουμε ανισότητες. Η Επιτροπή Φόντερ Λάιεν θέλει ε, να είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ε, κάνει προσπάθειες για παραπάνω. Για τη γενιά μας η Ευρώπη είναι ένα όραμα το οποίο ε, δημιουργήθηκε για να φέρει ειρήνη, ευημερία και ενότητα. Για τα παιδιά μας η Ευρώπη πρέπει να είναι κάτι πολύ περισσότερα. Μας λένε πολύ δυνατά και ξεκάθαρα ότι υπάρχει μεγάλη επιθυμία να ζουν σε ένα φυσικό και υγιή ε, πλανήτη με πράσινο και βιώσιμη ε, ανάπτυξη. Εγώ έχω αφιερώσει τη ζωή μου στα δημόσια αξιώματα. Έχω εκλεγεί τρεις φορές στο Εθνικό Κοινοβούλιο μου και είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχω περάσει 27 χρόνια να εργάζομαι με παιδιά και εφήβους ως κλινική ψυχολόγος σε δημόσια νοσοκομεία για θέματα ψυχικής υγείας, για αυτούς που ξεχνάμε πολύ συχνά. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τη σημασία των συστημάτων υγείας που λειτουργούν αποτελεσματικά και η συλλογική υγεία της κοινωνίας μας εξαρτάται από την ατομική υγεία κάθε πολίτη. Αυτό όμως δεν αρκεί από μόνο του. Εξαρτάται και από τη γενικότερη υγεία του πλανήτη μας. Βρίσκομαι λοιπόν ενώπιόν σας σήμερα προκειμένου να αφιερώσω όλη μου την ενέργεια, όλες μου τις γνώσεις και όλες μου τις ικανότητες για να υπηρετήσω αυτούς τους ευρωπαϊκούς σκοπούς ως Επίτροπος Υγείας για την επόμενη πενταετία. Αγαπητοί φίλοι, η υγεία είναι ένας τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει προσπάθεια για περισσότερα. Δεν μπορούμε να παβόμαστε σαν όσα έχουμε επιτύχει. Υπάρχουν αλλαγές στο κλίμα, στην τεχνολογία και δημογραφικές αλλαγές, οι οποίες αλλάζουν την κοινωνία μας και τον τρόπο ζωής μας. Η Ευρώπη πρέπει να έχει τα ενία της μετάβασης σε ένα πιο υγιεινή πλανήτη και σε ένα νέο ψηφιακό κόσμο. Αυτές είναι προκλήσεις οι οποίες όλες έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα ζωή μας, έχουν αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, στην ανταγωνιστικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη. Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά με, αν έχουμε μία προσέγγιση που ε, βάζει την υγεία στην πρώτη γραμμή. Μία υγεία και υγεία σε όλες τις πολιτικές. Η Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal, είναι μία ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις ολιστικά. Θέτει την καλή υγεία, τη βιώσιμη, τη διατροφή, τα τρόφιμα τα οποία μπορούμε όλοι να αγοράσουμε στην ίδια πολιτική ομπρέλα. Είμαι ικανοποιημένη που η δουλειά μου για την ασφάλεια των τροφίμων, την ευημερία των ζώων και την υγεία των φυτών θα είναι σημαντικό τμήμα αυτού του θεματολογίου και είμαι ενθουσιασμένη να ηγηθώ τη στρατηγική για μια νέα στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο για βιώσιμα τρόφιμα. Θα λάβω υπόψη μου κάθε τμήμα τη διατροφική αλυσίδα. Θα έρθω σε επαφή με κάθε φορέα και θα θέσω την κοινωνική ένταξη στο επίκεντρο. Αυτέ είναι οι προκλήσει που αναγνωρίζω αλλά δεν φοβάμαι να τις αντιμετωπίσω, διότι γνωρίζω ότι εσείς θα είστε βασικός εταίρος σε αυτή τη διαδικασία. Ως βουλευτής και εγώ ίδια αναγνωρίζω τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξαν αυτές οι επιτροπές και προσβλέπω στη στενή συνεργασία μαζί σας τα επόμενα χρόνια. Έχω συναντήσει πολλούς από εσά τις περασμένες εβδομάδες και μου είναι σαφές ότι έχουμε κοινέ απόψεις για πολλά θέματα. Το να προστατεύσουμε τους πολίτες από κινδύνους όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Το να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα φυτοφάρμακα. Το να προωθήσουμε την υγεία των ζώων και την ευημερία των ζώων. Αυτά είναι θέματα όπου θέλω να παλέψουμε μαζί. Παράλληλα, θα δουλέψω στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σε αυτό το τομέα είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί αντιπεραιτέρω. Είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε τη ζημιά που γίνεται στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη δημόσια υγεία όταν δεν εφαρμόζονται οι κανόνες. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνη είναι επιτακτική ανάγκη αν θέλουμε να επιτύχουμε. Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια πρέπει να είναι η φάρη στην προσπάθεια. Πρέπει να σταματήσει η απάτη στα τρόφιμα που υποσκάπτει την ενιαία αγορά και την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Θέλω να εξασφαλίσω ότι έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να διατηρήσουμε υγιείς τους πολίτες μας και γι' αυτό χρειάζεται μια σταθερή ροή προσιτών φαρμάκων. Το φαρμακευτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δώσει στους πολίτες υψηλής ποιότητας και προσιτά φάρμακα για δεκαετίες. Θα εστιάσω στην εφαρμογή ενός εξυγχρονισμένου και πιο στεναρού νομοθετικού πλαισίου για τις ιατρικές συσκευές. Αυτό πρέπει να γίνει ούτως ώστε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των ασθενών και να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα αυτό. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην προσπάθεια αυτή, γιατί μπορεί να φέρουν συγκεκριμένα ωφέλη σε ασθενείς και στου επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Θέλω να ενισχύσω αυτό το δυναμικό και θεωρώ ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για όλα αυτά τα θέματα η Ευρώπη μπορεί να παίξει έναν ειδικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αγωνίζεται για περισσότερα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ομφαλοσκοπεί. Η εμβέλεια των δράσεών μα θα πρέπει να είναι παγκόσμια και πολυμερή και να ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορά μα. Η μικροβιακή αντοχή είναι ένα κίνδυνο που αφορά την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Ο χρόνος περνάει και πρέπει να δράσουμε τώρα. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προπομπός στην παγκόσμια προσπάθεια και εγώ είμαι υπέρ μιας διεθνούς συμφωνίας για τη χρήση και την πρόσβαση στα αντιμικροβιακά φάρμακα. Για αυτό το λόγο δίνω προτεραιότητα στην εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αντίληψης για την υγεία εναντίον της μικροβιακής αντοχής. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω με τον καρκίνο. Μια εμβληματική προτεραιότητα για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με αφορά και εμένα την ίδια πολύ προσωπικά. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την νίκη κατά του καρκίνου. 40% από εμά θα πάθουμε καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή μα. Δεν υπάρχουν πολλέ οικογένειε που δεν έχουν κάποιον ο οποίο νόσησε από αυτή την αρρώστια. Αυτό από μόνο του είναι λόγο ούτω ώστε να βάλουμε τον καρκίνο πάνω-πάνω στι προτεραιότητέ μα στον τομέα τη υγεία. Το να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο και να νικήσουμε τον καρκίνο απαιτεί όλου και την προσπάθεια όλων και μια πραγματικά οριζόντια προσέγγιση όπου θα εντάσσει την υγεία σε όλες τις πολιτικές. Τα πάντα, από τα τρόφιμα που τρώμε, τη ζωή που κάνουμε, τα φάρμακα, την περίθαλψη, την τεχνολογία στην οποία έχουμε πρόσβαση, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να νικήσουμε τον καρκίνο. Καθένα από αυτά είναι ένα κρίκο σε μια λυσίδα που έχει ένα μόνο στόχο, να μειώσει την επίπτωση του καρκίνου στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι το σχέδιό μας το να νικήσουμε τον καρκίνο, ότι αφορά όλες τις δράσεις που υπάρχουν στην επιστολή μου για την αποστολή μου. Από τη στρατηγική, από το χωράφι στο πιάτο, την πράσινη συμφωνία, τη μικροβιακή αντοχή, την φθηνή καινοτομία των φαρμάκων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόληψη, τη διάγνωση, την θεραπεία, την έρευνα, τη ζωή μετά τον καρκίνο και την ανακουφιστική και παρηγορητική αγωγή. Πρέπει να εμπλέξει τομεί και κλάδου πέρα από το τομέα τη υγεία, συμπεριλαμβάνοντα την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Έχω συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον καρκίνο στο παρελθόν ω πρόεδρο του Europa Donna, μια, ένας ευρωπαϊκός για τον καρκίνο του στήθους. Ε, ως σύμβουλος των ασθενών, σε συνεργασία με του γιατρούς, τον κλάδο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια. Ήμουν μία από αυτούς που ανεπλάκησαν στο να υιοθετηθεί το πρώτο ψηφίσμα για τον καρκίνο του στήθους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2003. Το να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των ασθενών που έχουν νοσήσει από καρκίνο ήταν πάντα μία από τις βασικές μου αρχές. Και μιλάω από προσωπικέ εμπειρίες. Σας διαβεβαιώ λοιπόν γι' αυτό ότι θα συνεχίσω αυτές τις αρχές να τις χρησιμοποιώ στην τρέχουσα αποστολή μου, εάν με επιβεβαιώσετε ω Επίτροπο. Κυρίε και κύριοι, αν γίνω επίτροπο, αυτό θα μου δώσει τη δύναμη και την ευκαιρία να στρίξω αρχές τις οποίες πίστευα και για τις οποίες πολέμησα με πάθος όλη μου τη ζωή. Θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα κράτη-μέλη, με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με τους συναδέλφους μου επιτρόπους για να βελτιώσω τη δημόσια υγεία και να εξασφαλίσω ένα βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη. Όταν εντοπίζουμε αδυναμίες στα συστήματά μας, θα πρέπει από κοινού να βρούμε και τη θεραπεία, να δουλέψουμε με ζήλο, φιλοδοξία και δέσμευση. Το να στήσουμε και να οικοδομήσουμε εταιρικέ σχέσεις που να βασίζονται στην ειλικρίνεια, τιμιότητα, διαφάνεια και λογοδοσία είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί από εσά με ρωτήσατε στο Στρασβούργο τι ελπίζω να πετύχω με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το σκεφτόμουν λοιπόν, θα σας πω, από την πρώτη μέρα αυτού του ταξιδιού. Σε πέντε χρόνια μετά από πέντε χρόνια, θέλω όλοι μαζί να κοιτάξουμε προ τα πίσω και να πούμε υιοθετήσαμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον καρκίνο και μειώσαμε τον πόνο που προκαλεί ο καρκίνο. Έχουμε δώσει πιο υγιή και πιο πράσινα τρόφιμα στου πολίτε μα. Βελτιώσαμε τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση των ασθενών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αγγίξαμε τις, ε, την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Εξασφαλίσαμε ότι η Ευρώπη δουλεύει για όλου του πολίτε στον τομέα τη υγεία. Αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις και δώσαμε αποτελέσματα. Γι' αυτό είμαι εδώ ενώπιόν σας σήμερα για να ζητήσω τη στήριξή σας για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους μαζί. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις για να εμπνεύσουμε, για να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας προς τις μελλοντικές γενιές. Εν τη ενώση ισχύς. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα οργανωτικά. Εφτά ερωτήσεις για κάθε μία από τις ε, πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ερωτήσεις από τους συντονιστές ή τους εκπροσώπους τους και στη συνέχεια έχουμε 18 ερωτήσεις οι οποίες ε, ε, θα γίνουν βάση του κανόνα DON'T και επισημαίνω ότι θα υπάρχουν και ερωτήσεις οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα τεθούν και από τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας που είναι ε, συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη ακρόαση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη από τις επτά ερωτήσεις των επτά πολιτικών ομάδων ε, για το ΕΛΚ, η κυρία Ντολόρε Μοντσεράτ, για 1,5 λεπτό το πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Αντιπρόεδρε, υπο... Επίτροπε, ε, πραγματικά ταυτίστηκα με τα όσα είπατε για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ε, Όλοι μας νομίζω έχουμε ζωήσει τον καρκίνο από κοντά ή σε πρώτο πρόσωπο. Είναι μια ε, ασθένεια η οποία τίνει να γίνει η πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Πάνω από το 40% των Ευρωπαίων είπατε ότι ε, θα νοσήσουν από καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή τους. 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα χάσουν τη ζωή τους φέτος από καρκίνο. Οι ασθενείς ε, με καρκίνο στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχουν 30% ε, λιγότερες ε, πιθανότητες θεραπείες από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πέραν όμως της σκληρή πραγματικότητας υπάρχουν λόγοι για να ελπίζουμε. Η Ευρώπη έχει εξαιρετικούς επαγγελματίες και ερευνητές. Η θνησιμότητα έχει πέσει κατά 10%. Μεταξύ του 30% και 50% των καρκίνων είναι πλέον ε, θεραπεύσιμοι και μπορούν να αποφευχθούν. Εάν επενδύσουμε περισσότερα λοιπόν στην πρόληψη και αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε την πρόορη διάγνωση θα μπορέσουμε να ε, διπλασιάσουμε τα ποσοστά επιβίωσης. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, εμείς στο ΕΛΚ ε, έχουμε τα ενία στο σχέδιο της Ευρώπης για την καταπολέμηση του καρκίνου και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον θα έχετε μέτρα για να ε, εγγυηθείτε την ισότητα στην πρόσβαση για τις θεραπείες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μονσεράτ για αυτή την ερώτηση. Πράγματι, όπως σας είπα, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο με αγγίζει ιδιαίτερα προσωπικά. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου πρέπει να καλύψει όλα όσα αναφέρατε. Και αυτό το σχέδιο, αν όντω αποβεί αποτελεσματικό, δεν μπορεί να αφήσει κανέναν πίσω. Δεν μπορούμε να μιλούμε για ανισότητε όταν συζητούμε τη θεραπεία για τον καρκίνο και τη φροντίδα για τον καρκίνο. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε όλε τι πτυχέ από την πρόληψη στην παρηγορητική αγωγή, διότι πραγματικά είναι απαράδεκτο όταν γνωρίζουμε σήμερα ότι μπορεί να προληφθούν περίπου 30% όλων των μορφών καρκίνου, να μην επενδύουμε αρκετά για να αλλάξουμε τρόπο ζωής, το οποίο γνωρίζουμε ότι θα, βελτιώ, ε, θα βελτιώσει την κατάσταση και θα οδηγήσει σε λιγότερο πόνο. Θα ήθελα να αναφέρω και κάτι που είπατε κι εσείς για τη διάγνωση. Πολλές χώρες έχουν ε, προγράμματα ε, διάγνωσης, αλλά για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα και πρέπει να ακολουθούν ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. Και γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, το 2019 πέρασε ένα ψήφισμα για τους ε, καρκίνους των γυναικών ε, και τον ε, ιό HPV. Η πρόσβαση στα φάρμακα, προσιτά φάρμακα, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου και αυτό φυσικά θα συμβαδίζει και με άλλες πτυχές τις οποίες πρέπει να εξετάσουμε και τις οποίες ανέφερα. Ανέφερα στην αρχική μου παρέμβαση τον ε, κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής. Πολλοί ασθενείς που νοσούν από καρκίνο χάνουν τη ζωή τους ακριβώς λόγω της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Πρέπει να δούμε λοιπόν το πρόβλημα οριζόντια και να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ε, σε όλες τις πολιτικές για την υγεία και όχι μεμονωμένα στο περιθώριο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ε, μεγάλο χρόνο ε, από την ε, δουλειά μου. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, Πρέπει να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους Ευρωπαίους ασθενείς. Ε, δεν θα πρέπει κανείς να μείνει πίσω στη μάχη κατά του καρκίνου. Δεν πρέπει να υπάρχουν ε, ε, ασθενείς πρώτης και δεύτερης γραμμής της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες συνεργασίες και πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα αυτή της Βαλέτα, του Λουξά. Ήταν θετικέ προσπάθειες, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Σας προτείνω λοιπόν από κοινού να προωθήσουμε μια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει ίση πρόσβαση τη θεραπεία και να έχουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση του καρκίνου αλλά και όλων των ασθενειών. Ο καρκίνο έχει πολλά πρόσωπα και θα πρέπει να ασχοληθούμε με όλα αυτά. Επίση, θα πρέπει να βελτιώσουμε ε, την προσοχή προ του ασθενεί, να είναι ολιστική όπω είπατε και εσεί και να μην αφορά μόνο την ιατρική πτυχή αλλά και την κοινωνική βοήθεια προ του ασθενεί και τα μέλη τη οικογένειά του. Και επίση και την ψυχική υγεία τη κοινωνία μα. Το άγχο, η κατάθλιψη, ε, το στρες ε, όλα αυτά είναι ε, ε, στοιχεία που απαιτούν να επενδύσουμε περισσότερο και να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τον καρκίνο. Τι μέτρα σκοπεύετε να προωθήσετε για να βελτιώσετε τις επενδύσεις στην έρευνα κατά του καρκίνου. Συγγνώμη, πριν απαντήσετε, σας παρακαλώ να τηρείτε την έννοια της συμπληρωματικής ερώτησης 45 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ. το σχέδιο να νικήσουμε τον καρκίνο της Ευρώπης ασχολείται με όλα. Είπατε ότι υπάρχουν ανισότητες στην πρόσβαση στη θεραπεία. Εγώ να σας πω κάτι θετικό που προέκυψε από τη δράση του Κοινοβουλίου. Είναι η οδηγία για την δια συνοριακή υγεία. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν συνεργαζόμεθα μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή των ασθενών. Επίσης υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς. Δίνει πρόσβαση σε στοιχεία για παιδικές ασθένειες, για σπάνιες ασθένειες και άλλες σπάνιες μορφές καρκίνου, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ο ασθενής. Πιστεύω στη συνεργασία μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν έχω βέβαια μια ταχεία απάντηση σε όλα για την έλλειψη φαρμάκων, για παράδειγμα. Είπα ότι αν επιβεβαιωθώ θα δεσμευθώ για να προωθεί το σχέδιο να νικήσουμε τον καρκίνο. Ευχαριστώ. Για τη σοσιαλιστική ομάδα, ο κύριος Γκουτάλαντ. Η κυρία Γκουτάλαντ. Η έκθεση, ακόμα και σε χαμηλές δόσεις ενδοκρινικών διαταρακτών, οδηγεί σε πολύ σοβαρές αρρώστιες όπως ε, καρκίνος, διαβήτης, ε, έλλειψη γονιμότητα και άλλε αρρώστιε. Και ειδικά τα μικρά παιδιά είναι πολύ ευαίσθητα. Πέρα από τον ανθρώπινο πόνο, αυτά τα πράγματα κοστίζουν και πάρα πολύ. Πάνω από 160 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω είναι το κόστο αυτό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν οι άνθρωποι να αποφύγουν αυτέ τι ουσίε στην καθημερινότητά του, Γιατί υπάρχουν παντού. Στο νερό που πίνουμε, στα καλλιντικά, στα παιχνίδια, στι συσκευασίε των τροφίμων. Όλοι έχουν το δικαίωμα σε μια ζωή χωρίς να εκτίθονται σε αυτές τις ουσίες. Θα Πρόκειται να προτείνεται χωρίς ε, καθυστέρηση οριζόντια κριτήρια για να εντοπίζουμε αυτού του διαταράκτε σε όλου του τομεί. Μπορείτε να μα υποσχεθείτε σήμερα ότι θα αντιδράσετε με συγκεκριμένο τρόπο απέναντι σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα, αντί να κρύβεστε πίσω από την πολύ αδύνατη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρονολογείται από το 2018 ή πέρα από αόριστες ε, υποσχέσεις για το fitness check. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να βλέπω προ τα μπρό. Εγώ θα σχολιάσω για αυτά που θα ήθελα να κάνω, κυρία Γκούτλαντ, ε, στο μέλλον. Και σα ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτε είναι και στην επιστολή ανάληψη καθηκόντων. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι προτεραιότητα. Έχετε απόλυτα δίκιο. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Γιατί έχουν επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Αυτό είναι αναμφίβολο πλέον. Γνωρίζω το ψήφισμα του Κοινοβουλίου το φετινό, γνωρίζω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει πριν το 2020 να εγκριθεί νομοθεσία από αυτού. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα, να καθορίσουμε οριζόντια κριτήρια. Αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα. Έχει σημειωθεί πρόοδο τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν θέλω να πω πως δεν έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα, πολύ περισσότερα. Γιατί ξέρουμε ότι ο μόνος λόγος που εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον ω υποψήφια Επίτροπος Υγείας είμαι εδώ, ο μόνος λόγος είναι να δεσμευθώ να προστατεύσω του συμπολίτε μας και το περιβάλλον. Να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπατε. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για να δούμε το αποτέλεσμα της έκθεσης σε πολλαπλούς διαταράκτες και ουσίες. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα αυτό. Θα περιμένω να έχω τα αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας. Ήδη κάποια κράτη-μέλη έχουν σχέδια δράση για τα θέματα αυτά. Πρέπει να τα στηρίξουμε. Και πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι διαταράκτες αυτοί θα είναι ένα σημαντικό τμήμα των προτεραιοτήτων της επόμενης Επιτροπής. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Τώρα δεν θα ξεκινήσω συζήτηση μαζί σας για το θέμα αυτό, αλλά μία περαιτέρω διευκρίνηση. Συμφωνείτε ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι όσο επικίνδυνοι και ο ίδιος ο καρκίνος και άλλες ε, τοξικές ουσίες. Και είπατε ότι θέλετε μία διατομιακή προσέγγιση. Τότε πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ των ουσιών που θεωρούμε ότι είναι ύποπτες ω διαταράκτε και ήδη καλύπτονται και άλλες τοξικές ουσίε που δεν καλύπτονται ακόμη. Φυσικά και ούτε εγώ θέλω να ξεκινήσω συζήτηση μαζί σας. Αυτό που θέλω, να, θέλω να έχουμε την ευκαιρία να ακούσω από εσά για να λάβω υπόψη όλες τις ανησυχίες σας. Γι' αυτό είπα ότι είμαι διαθέσιμη για να σας ακούσω. Τώρα δεν θα ήθελα να συγκρίνω την επικινδυνότητα των διαταρακτών αυτών με την επικινδυνότητα του καρκίνου, αλλά ξέρω ότι έχουν επίπτωση στην ε, υγεία των συμπολιτών μας, άρα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό δεσμεύομαι να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Αναμένουμε το τεστ καταλληλότητας και φυσικά προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το θέμα. Είμαι σαφής επί αυτού. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα ο λόγος... Σε μένα τον ίδιο. Θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου. Σωστό δεν είναι να μπορώ και εγώ να δώσω το λόγο στον εαυτό μου. Θα προεδρεύσει λοιπόν για ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα πρώην αντιπρόεδρος. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα για τα φυτοφάρμακα. Είπατε στην, απάντηση, στην γραπτή σας απάντηση στις δικές μας ερωτήσεις ότι πιστεύω ότι θα πρέπει από κοινού να σκεφτούμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε έναν υποχρεωτικό στόχο μείωσης του κινδύνου ε, στα, που συνδέεται με τα φυτοφάρμακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι από κοινού θα πρέπει να σκεφτούμε τη δυνατότητα που έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισοδυναμεί με το θα δράσουμε. Εξού και ένα απλό ερώτημα. Στα πλαίσια της στρατηγικής, από το χωράφι στο πιάτο, θα στηρίξετε ένα στόχο με νούμερα για τη μείωση των φυτοφαρμάκων και τον κίνδυνο που συνδέεται με τα φυτοφάρμακα ή όχι. Thank you Ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ισχυρή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα. Επίσης γνωρίζουμε ότι δεν εφαρμόζεται σωστά. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δημιούργησε την Επιτροπή ΠΕΣΤ, η οποία έδωσε σημαντικά αποτελέσματα και ήταν πολύ επικριτική για τα κράτη-μέλη, από ό,τι ξέρω. Η η έκθεση της Επιτροπής ζητάει διαφάνεια και λογοδοσία. Για μένα είναι πολύ σημαντική λέξη αυτή, η λογοδοσία. Γίνεται μια αξιολόγηση μέσω του refit που δεν έχει τελειώσει και θα πρέπει να την εξετάσουμε. Και ελπίζω και είμαι αισιόδοξη ότι οι αλλαγέ στη Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα θα, που θα συμπεριλάβει την διαφάνεια και αυτό θα είναι πολύ θετικό. Αυτό που μπορώ να πω, κυρία Καμφά, είναι το εξής. Ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεσμεύομαι για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα φυτοφάρμακα και να προσπαθήσουμε να επενδύσουμε και να ενθαρρύνουμε την εξέβρεση άλλων λύσεων χαμηλού κινδύνου. Αυτή είναι ευθύνη μας. Είναι τμήμα της ε, επιστολής ανάληψης των καθηκόντων μας και για την ε, Πράσινη Συμφωνία και για τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο. Θα το παρακολουθήσω εκ του σύνεγγυς, ούτως ώστε να δώσω αποτελέσματα. Ξέρω ότι οι πολίτες ανησυχούν, πρέπει να το σεβαστούμε αυτό και πρέπει να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε. τα φυτοφάρμακα έχουν επίπτωση στους ανθρώπους. Εξού και η ανάγκη να έχουμε έναν στόχο με νούμερα για τη μείωση. Αλλά να δούμε και τι επιπτώσεις έχει αυτό στις μέλισσες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε σε στη φάση απόρριψης της πρότασης της Κομισιόν για τη μέθοδο αξιολόγησης της επίπτωσης των φυτοφαρμάκων στις μέλισσες. Αν το Κοινοβούλιο σε λίγες εβδομάδες έχει αντίρρηση και δεν επικυρώσει την ε, τρέχουσα πρόταση της Κομισιόν, δεσμεύεστε εσείς ενώπιόν μας να δώσετε συνέχεια στις προτάσεις της ΕΦΣΑ, να ακολουθήσετε τα επιστημονικά στοιχεία και από κοινού εσείς και εμείς να πιέσουμε τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να δεχτούν τη σύσταση της ΕΦΣΑ να γίνει μια πλήρης αξιολόγηση της επίπτωσης των φυτοφαρμάκων στις μέλισσες. Μπορώ να δεσμευτώ στο εξή. στο βαθμό που μπορώ να δεσμευτώ ως υποψήφια επίτροπος, είναι ότι δεν θα χαμηλώσουμε τον πύχη στην προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η προστασία των μελισσών θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των πολιτικών μας και είναι και τμήμα της α, Πράσινης Συμφωνίας που αναφέρεται στην επιστολή ανάληψη των καθηκόντων μου. Γνωρίζω ότι το 2013, αν δεν κάνω λάθο, η Κομισιόν απαγόρευσε τρία νεονικοτινοειδή. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν σοβαρότατες δυσκολίες στην εφαρμογή του εγγράφου, του κατευθυντηρίου εγγράφου της ΕΦΣΑ για τις μέλισσες. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να εξετάσουν τώρα την οξία τοξικότητα, επανεξετάζουν τα αποτελέσματα, γιατί πρέπει να δούμε και τη χρόνια τοξικότητα και πρέπει να βρούμε συνένεση. Από πλευράς μου, η μείωση της χρήσης των νεονικοτινοειδών και η εξέβρεση εναλλακτικών λύσεων είναι πρώτη προτεραιότητα. Εργάζομαι όμως με βάση τη συνένεση και θα προσπαθήσω να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα κράτη-μέλη, για να βρούμε έναν τρόπο, ούτω ώστε να εφαρμόσουμε το κατευθυντήριο έγγραφο για τις μέλισσες, ούτω ώστε να μπορούμε να προστατεύουμε το περιβάλλον μας. Όταν μιλάμε για τις μέλισσες και τους επικονιαστές και ξέρω ότι στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου μου ε, υπάρχει ένα στοιχείο που είναι η, η δημόσια υγεία. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι λάθος. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση. Η υγεία είναι το φαγητό, είναι το περιβάλλον, είναι τα πάντα. Ε, και αυτά που είπε η κυρία Μονσεράτ πριν από λίγο. Όλοι ζούμε σε αυτό τον πλανήτη. Όλοι είμαστε τμήμα αυτού του πλανήτη και όλοι πρέπει να τον προστατεύσουμε. Και αυτό είναι δική μου ευθύνη. Ευχαριστώ. Ο... Η Μισελ Ριβαζή, εξ ονόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ και καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την απάντησή σας στον κύριο Καμφάν, διότι λέτε ότι η νέα Επιτροπή δεσμεύεται να επιτύχει το στόχο της μηδενικής ρήπανσης. Και ξέρετε ότι είχαμε πάρα πολλές ε, ε, συγκρούσεις ε, με τον προκάτοχό σας για τα φυτοφάρμακα, κυρίως για, το γλυφοσάτ, για Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγγνώμη, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα θέματα των φυτοφαρμάκων, σύστησε και ιδιαίτερη επιτροπή για τα θέματα αυτά και η παρούσα ε, επιτροπή δυστυχώς δεν έτεινε δίκον στα όσα είχε να πει η επιτροπή και ε, εμείς ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, εγκρίνει τις, ε, τους προσανατολισμούς της ΕΦΣΑ για τις μέλωσες. Αυτό είναι ο νόμος κυρία μου. Επομένως, τα φυτοφάρμακα μπορούν να, γίνουν, να εγκριθούν μόνο αν δεν έχουν καμία τοξική συνέπεια για τις μέλισσες. Παρ' όλα αυτά, ε, τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, δεν το δέχονται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένε φορέ δεν αναλαμβάνει την πρωτοβουλία που θα έπρεπε. Και ακόμα και αν έχουμε εμεί ενστάσει για το θέμα αυτό. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, εάν εσεί γίνετε επίτροπο, θα αλλάξετε τη στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προτείνετε μέσα στο επόμενο τρίμηνο ένα νόμο που θα λαμβάνει υπόψη τι συστάσει τη ΕΦΣΑ για τη χρόνια τοξικότητα η οποία προβλέπεται στην νομοθεσία για τι μέλη Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση ε, αντιλήφθηκα και την απογοήτευσή σας, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω για ό,τι έχει συμβεί. Αυτό στο οποίο μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι εμείς βλέπουμε το θέμα με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει συγκεκριμένο ε, αναφορά στο θέμα στην επιστολή της αποστολής μου και τι υπάρχει και πρόβλεψη της ε, Προέδρου. Και υπάρχουν προτεραιότητες ε, για τα φυτοφάρμακα. Εγώ είμαι βουλευτής. Η νομοθεσία ε, ε, ψηφίζεται για να εφαρμόζεται και όλοι αυτό πρέπει να κάνουμε. Να προωθούμε αυτό. Με ρωτήσατε λοιπόν αν δεσμεύομαι να προωθήσω νομοθεσία εντός τριών μηνών. Γνωρίζετε ότι εργαζόμαστε ως σύνολο το Σώμα των Επιτρόπων, αλλά μπορώ να δεσμευτώ ως προς το εξή. Μπορώ να δεσμευτώ ότι θα προσπαθήσω να βρω την κατάλληλη συνένεση προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για να υπάρχει εφαρμογή της νομοθεσίας. Και εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι αυτά είναι απλώς ε, κενά λόγια. Είναι τμήμα της εντολής μου. Το, από το χωράφι στο τραπέζι είναι τμήμα της εντολής μου. Η εφαρμογή του Green Deal που είναι και αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου Τίμερμανς είναι η εντολή μου. Και πρέπει να συνεργαστώ με όλους προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα. Αναγνωρίζω και νομίζω ότι αναγνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχει εφαρμοστεί καταλήλω νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα. Η Επιτροπή ΠΕΣΤ ε, είχε μια έκθεση η οποία ήταν ιδιαίτερα επικριτική και σας ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά είπε και αλήθειες. Και τώρα ε, τα πράγματα είναι ε, στα χέρια της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν εγώ επιβεβαιωθώ ως Επίτροπος θα προσπαθήσω να προωθήσω το θέμα αυτό απαντάτε, αλλά όχι ακριβώς ε, στην ερώτησή μου. Διότι το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ο νόμος του 2009, ο οποίος απαιτεί να λάβουμε υπόψη τις χρόνιες συνέπειες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δεν το σέβονται αυτό. Εγώ λοιπόν σας ζητώ να προτείνετε μια νομοθετική πράξη στο Συμβούλιο. Πρέπει να κάνετε κάτι ε, το οποίο θα είναι σε πολιτικό επίπεδο και όχι σε τεχνικό επίπεδο. Αν υπάρχει λοιπόν κάτι σε πολιτικό επίπεδο και υπάρχει ειδική πλειοψηφία θα μπορέσουμε και εμείς ως Κοινοβούλιο να δράσουμε απέναντι στα κράτη-μέλη. Αν δεν έχετε στήσει το να προτείνετε νόμο στο Συμβούλιο, μια νομοθετική πράξη, ε, τι θα κάνετε. Και αν γίνετε επίτροπος θα κάνετε την κατάλληλη πρόταση για να λάβετε υπόψη τους προσανατολισμούς της ΕΦΣΑ για τις μέλεσες και, τις, ε, και να γίνουν αυτά σε επίπεδο Συμβουλίου, να είναι σε πολιτικό επίπεδο και όχι σε τεχνικό επίπεδο. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν είναι τεχνικής φύσεως. Γι' αυτό και ακριβώς προηγουμένως είπα ότι θα ήθελα να μου δοθεί ευκαιρία να συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη και να το προωθήσω το θέμα αυτό, διότι έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούμε να βλέπουμε απλώς την οξία τοξικότητα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα για να δούμε τη χρόνια τοξικότητα και εγώ θα βασιστώ στις επιστημονικές ενδείξεις. Αυτό για το οποίο δεσμεύομαι είναι ότι θα ασχοληθώ με το θέμα και θα το προωθήσω για έναν και μόνο λόγο, διότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σκέλος της προστασίας του πλανήτη μας, του περιβάλλοντός μας και της καθημερινής μας ζωής εντός του Green Deal, της Πράσινης Συμφωνίας και της πρότασης για το χωράφι στο τραπέζι. Ευχαριστώ. Εξαρτησία και δημοκρατία. Σιλβία Νίνερ. Λοιπόν, διάβασα πολύ προσεκτικά τις ε, γραπτές σας απαντήσεις. Και γι' αυτό θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις που δεν έχουν ε, να με αυτές τις γενικολογίες για βιωσιμότητα κτλ. Για παράδειγμα, για τους δωρητές οργάνων. Στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για αυτά. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή υπάρχει ο λεγόμενος κανονισμός αντίρρησης. Ερώτηση λοιπόν. Εσείς θέλετε να διατηρήσετε τις αρχές της επικουρικότητας με βάση τις οποίες ε, κάθε κράτος μέλος καθορίζει τους ε, κανόνες ε, μόνο του. Ή θέλετε να εισαγάγετε ένα ενιαίο σύστημα. Και πώς θα έπρεπε να είναι αυτό το σύστημα. Γιατί όπως ξέρετε χρειάζεται έγκριση για να υπάρξει παροχή οργάνων. Επίσης μιλήσατε για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Αλλά δεν ασχοληθήκατε με ένα πολύ βασικό θέμα. Ότι δεν ε, αναπτύσσονται νέε ενεργέ ουσίε. Πώ θέλετε να βοηθήσετε την έρευνα και ανάπτυξη, όταν είναι πολύ ψηλό το κόστο για να μπει στην αγορά ένα νέο αντιβιωτικό. Αυτά τα λεγόμενα αντιβιωτικά τελευταία καταφυγή και μετά δεν χρησιμοποιούνται. Άρα δεν αξίζει πλέον για τι φαρμακομηχανίε να τα αναπτύξουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα επιχειρήσω να απαντήσω στην ερώτηση, στις δύο ερωτήσεις για τις οποίες ευχαριστώ σε δύο λεπτά. Τώρα, δόρηση οργάνων. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για τα κράτη-μέλη, γιατί ξέρουμε ότι εξαρτάται η επιβίωση πολλών συμπολιτών μας από αυτό. Οπότε, προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφάλεια. Πρέπει να στηρίξουμε την καινοτομία γιατί πρέπει να γίνουν περισσότερα για το θέμα αυτό. Γνωρίζω ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει δυνατότητα κάποιο να ζητήσει να εξαιρεθεί από αυτό το σύστημα. Αλλά αυτό δεν έχει λειτουργήσει σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίση γνωρίζω ότι υπάρχει μια αξιολόγηση που επίκειται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του χρόνου νομίζω. Οπότε θα περιμένω να τη δω πριν αποφασίσω τι περαιτέρω πρέπει να γίνει. Τα κράτη-μέλη έχουν προγράμματα δράση, αλλά αν χρειάζεται τώρα μια ευρωπαϊκή στρατηγική, θα περιμένω να δω την αξιολόγηση. Αναγνωρίζω ότι είναι μεγάλη σημασία το θέμα, διότι έχει να κάνει με τόσα άτομα και υπάρχουν τόσα άτομα στις λίστες αναμονής για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Έχετε δίκιο. Δεν ανέφερα τι θα κάνουμε για αυτό το θέμα. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα έχουμε 30.000 ε, θανάτους στην Ένωση λόγω αυτού του φαινομένου το χρόνο. Το 2017 υπήρχε το δεύτερο πρόγραμμα δράσης τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν δεν κάνω λάθο, ίσως και να κάνω λάθος, υπήρχαν 70 ε, δράσεις ε, με βάση το θεματολόγιο για μία υγεία, στόχο του οποίου είναι να αντιμετωπίζουμε από κοινού τα άτομα τα ε, ζώα και το περιβάλλον. Βεβαίω χρειάζεται συνολική απάντηση. Γι' αυτό ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και το G20 ασχολούνται με το θέμα αυτό και τμήμα αυτή τη προσπάθεια είναι να ενθαρρύνουμε τον κλάδο μέσω καινοτομία να μα δώσει νέα αντιβιωτικά. Είναι, είναι πρόβλημα με ολέθριες συνέπειες, ε, δεν σταματάει στα σύνορα, πρέπει να υπάρξει συνολική απάντηση. Εγώ θα ήθελα η Ευρώπη να ηγείται αυτή τη προσπαθία. Ναι, αλλά δεν απαντήσατε καμία ερώτησή μου. Πρώτον, σας ρώτησα ποια είναι η προσωπική σας άποψη. Εάν για σας χρειάζεται ένας κανονισμός για τους δωρητές οργάνων, εσείς το αποφύγατε. Αλλά αυτό δεν με εξαφνιάζει. Επίσης, για την αντίσταση σε αντιβιωτικά. Δεν αναφέρατε το πρόβλημα. Πώς θέλετε να προωθήσουμε νέα αντιβιωτικά αν αυτά τα λεγόμενα τελευταίες καταφυγής δεν χρησιμοποιούνται. Δεν απαντήσατε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να απαντήσετε. Ναι, ήταν ερώτηση. Αλλά κοιτάξτε, μπορώ να σας δώσω μόνο τις απαντήσεις ε, στις οποίες ειλικρινά πιστεύω. Αν θα υπάρξει μια συνολική στρατηγική για την Ευρώπη για τους δωρητές οργάνων, θα ήθελα πρώτα να δω την αξιολόγηση. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα την έχουμε. Ούτω ώστε να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση, πώς μπορούμε να την αλλάξουμε. Με βάση στοιχεία, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία για να λάβουμε σωστές αποφάσεις. Πολύ εύκολα θα ήταν να σας πω τώρα, ναι βεβαίω, θα προτείνω μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν μπορώ να τεκμηριώσω. Να έχω επαρκή στοιχεία. Η αξιολόγηση της Κομισιόν θα βγει μέχρι το τέλος του χρόνου. Για την αντίσταση αντιβιωτικά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ηγέτε μέσω σωστών πρακτικών. Πρέπει να βοηθήσουμε τις φαρμακοβιομηχανίες με καινοτομία ούτω ώστε να προκύψουν νέα αντιβιωτικά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η Ευρώπη των μεταρρυθμιστών και ε, συντηρητικών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε απάντηση στα ερωτήματα που σας θέσαμε και που απαντήσατε γραπτώς, είπατε ότι η στενή συνεργασία με το Σώμα των Επιτρόπων και τους εκπροσώπους των άλλων ενδιαφερομένων φορέων και του κλάδου είναι σημαντικό για να υλοποιήσουμε τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είπατε ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη δημόσια υγεία, την έρευνα, την επιστήμη και την πολιτική για την υγεία. Αναφέρατε κάποιες προθέσεις για την ε, ολοκληρωτική κινητικότητα των ε, φορέων που εμπλέκονται. Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ε, DG Sante, τη DG DEFCO και την υπεύθυνη για την έρευνα Γενική Διεύθυνση και την απλούστευση των καθηκόντων τους στον τομέα της πολιτικής υγείας, ούτως ώστε, ούτως ώστε οι δράσεις να είναι πλήρεις και να ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο, ειδικά με το στόχο υπαριθμών 3. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πάντα μπορούμε να βελτιώνουμε τον συντονισμό. Η υποψήφια πρόεδρος είπε ξεκάθαρα το πώς θα συνεργαστούμε ως σώμα επιτρόπων και πολλοί από τους τομείς, ειδικά ο τομέας που μας απασχολεί σήμερα, η υγεία είναι ένας οριζόντιος τομέας. Εάν γίνω επίτροπος, το καθήκον μου θα είναι να συνεργαστώ με όλους τους υπόλοιπους επιτρόπους που ασχολούνται με την ε, στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο και με την πράσινη ε, συμφωνία, τον Επίτροπο Τίμερμανς, τον Επίτροπο Σχοινά και την ε, Επίτροπο Βεστάγκερ. Γιατί θα πρέπει το ψηφιακό θεματολόγιο να ενταχθεί στην πολιτική για την υγεία. Η πρόθεσή μου θα είναι να συνεργαστώ στενά με όλους, ούτω ώστε να δώσω αποτελέσματα. Αυτά ειδικά που υποσχέθηκα. Σε σχέση με τον καλύτερο συντονισμό, Εγώ συνεργάζομαι με όλους τους φορείς, με όλες τις οργανώσεις, προσπαθώ να χτίσω συνένεση, προσπαθώ να δω πού υπάρχουν εμπλοκές και δεν είναι απλά τα πράγματα και πώς μπορώ να βοηθήσω για να τα πλουστεύσουμε. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την προσέγγιση στα πλαίσια της εντολής μου, να ακούω προσεκτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους βουλευτές, που πολλές φορές βλέπουν κάτι που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Επομένως, λέω ναι. Θεωρώ ότι η στενή συνεργασία με τους άλλους επιτρόπους είναι επιτακτική ανάγκη. Θεωρώ ότι ο καλύτερος συντονισμός είναι απαραίτητος σε κάποιους τομείς και αυτά θα είναι τμήμα των δικών μου καθηκόντων εάν γίνω επίτροπος. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την μεταρρύθμιση και τον ανασχηματισμό και την αλλαγή των θεματολογίων των γενικών διευθύνσεων μπορεί να συνεισφέρει σε, στο να επανέλθει στην Ευρώπη η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, ούτως ώστε να είναι πιο ασφαλής η ήπειρός μας και παράλληλα να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα απαραίτητα φάρμακα. Ξέρω ότι αυτό απασχολεί πολλούς από εσά και ξέρω ότι εξαρτόμαστε από φάρμακα που έρχονται από τρίτες χώρες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γι' αυτό. Πρέπει να δούμε τι επίπεδα ελέγχου έχουμε για να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή αυτά τα φάρμακα. Φυσικά θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία και να επενδύσουμε σε αυτό και η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ηγέτης σε ό,τι αφορά την καινοτομία της φαρμακοβιομηχανίας. Είναι σημαντικό να το πετύχουμε αυτό. Όλο το πακέτο που συζητάμε σήμερα εμπλέκει και θέματα ψηφιοποίησης και πρέπει σίγουρα να παρακολουθούμε τις επιστημονικές εξελίξεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πολιτικές, όλους τους τομείς πολιτική. Επειδή έχω δουλέψει στον ε, τομέα της υγείας και επειδή είμαι και βουλευτής, είμαι σε επαφή με ανθρώπους που χρειάζονται φάρμακα συνεχώς. Και ξέρω τι σημαίνει να υπάρχει έλλειψη φαρμάκων, ξέρω τι σημαίνει να, υπάρχουν, να ε, υπάρχει πρόβλημα γιατί τα φάρμακα είναι πολύ ακριβά και όχι προσιτά. Μακάρι να ερχόμουν εδώ και σα έλεγα τσακ έχω την απάντηση. Αλλά δυστυχώ δεν την έχω. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα πρέπει να δούμε όλο τον τομέα, θα πρέπει να δούμε τι τιμέ και την επιστροφή των, των εξόδων. Υπάρχει μια νομική υποχρέωση τη φαρμακοβιομηχανία, ούτω ώστε να υπάρχει πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα. Πρέπει να συνεργαστούμε στενά και να έχουμε μια συνολική φαρμακευτική πολιτική για να υλοποιήσουμε αυτά που πρέπει να υλοποιήσουμε προ όφελο των ασθενών. Και κάτι που δεν αναφέρθηκε, ίσως αναφερθεί αργότερα. Η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και είναι ένα από τα βήματα που πρέπει να κάνουμε, εάν θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτά που λέμε. Θα το εξετάσω λοιπόν αυτό και ένα πιθανό νέο επιχειρηματικό μοντέλο, ούτως ώστε η Ευρώπη να είναι πολύ ψηλά να παίζει ηγετικό ρόλο στο θέμα αυτό. Κατε, Κατερίνα Κονιέσκα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, θα ήθελα να σταθώ στη τελευταία σας φράση που έχει σχέση και με την ερώτησή μου. Βάσει του Ευρωβαρομέτρου, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θα ήθελαν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχολείται περισσότερο με την υγεία και κάποιοι από αυτούς ε, φρονούν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα υγείας είναι ανεπαρκή. Είμαι βέβαιη ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς, όπως και εγώ, ότι φαίνεται ότι δεν έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι τα ίδια δικαιώματα πρόσβαση σε θεραπεία, το οποίο ισχύει για τις σπάνιε νόσους, αλλά όχι μόνο για τις σπάνιε νόσους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμβαθύνεται λόγω της έλλειψης ε, της κοινή ε, αξιολόγηση για τι τεχνολογίε τη υγεία. Είπατε ότι εάν ε, τα καταφέρετε, χρησιμοποιήστε τον όρο θα τα καταφέρετε, αλλά σκοπεύετε να προωθήσετε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία του. Τι θα κάνετε για να ε, βγούμε από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει το Συμβούλιο, διότι χωρί ε, την αξιολόγηση τη τεχνολογία υγεία δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά την πρόσβαση ε, ασθενών σε υπηρεσίες υγεία. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε το 2018 και νομίζω ότι υπήρχε και ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου το 2019, αν δεν κάνω λάθο. Η αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας είναι κομβική σημασία γιατί επιτρέπει στους ασθενείς να γνωρίζουν ε, εάν είναι ασφαλή τα φάρμακα τα οποία λαμβάνουν, αν ε, θα υπάρξει μία εξέταση για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για το κατά πόσον είναι ασφαλής και είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης γιατί επιτρέπει την καινοτομία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από πλευράς κρατών μελών ε, για να προχωρήσει το θέμα. Αλλά πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι καμία χώρα δεν θα πρέπει να μείνει πίσω. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους μας τους πόρους, πρέπει να υπάρχουν κοινά πρότυπα, προκειμένου να προστατεύσουμε τους ασθενείς. Και αυτό, κατά την άποψή μου, ε, είναι κάτι ε, το οποίο θα προσπαθήσω να επιτύχω με ιδιαίτερο στένος, να προσπαθήσω να έχω την απαραίτητη συνένεση, ώστε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018 που αφορά την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ε, να προχωρήσει. Διότι θεωρώ ότι είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα οποιοδήποτε συστήματος υγείας που θέλουμε να προωθήσουμε εμείς ως Ευρωπαίοι. θα ήθελα να σας πω ότι αυτό δεν αφορά μόνο την ασφάλεια, αλλά και την αποτελεσματικότητα. Η αναζήτηση συνένεσης και σας εύχομαι καλή τύχη στη συνένεση μεταξύ των κρατών μελών θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και οι συνάδελφοι ε, που θα με τα κράτη-μέλη ότι δύσκολα θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε υγεία για όλους και ασφάλεια για την υγεία για όλους. Στην ε, αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας καταφέραμε να συμπεριλάβουμε και τη διάσταση του ασθενούς. Ε, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον θα επεκτείνεται και το ρόλο των ασθενών σε όλη την υπόλοιπη νομοθεσία για την υγεία. Σκοπεύετε να του λάβετε σοβαρά υπόψη και να σεβαστείτε την άποψή τους. Πρόκειται για μια δύσκολη ερώτηση και θα την απαντήσω έτσι εν θερμό. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρμαχος των ασθενών. Είμαι υπέρμαχος των ασθενών διότι δεν είναι ίσως ε, γνωστό αλλά έχω διαγνωστεί και έχω περάσει θεραπεία για τον καρκίνο και έχω συνεργαστεί πάρα πολύ στενά με την κοινότητα των ασθενών και στη χώρα στην οποία ε, ζω έχουμε καταφέρει να έχουμε νομοθεσία που επιτρέπει στους συλλόγους ασθενών να έχουν μια θέση στο τραπέζι κάθε φορά που λαμβάνεται μια απόφαση που τους αφορά. Επομένω, απαντώ καταφατικά, θα συνεργαστώ πολύ στενά με του ασθενεί, αλλά θα συνεργαστώ στενά και με όλου του υπόλοιπου ενδιαφερομένους, προκειμένου να προσπαθώ να βρω τη σωστή άγουσα για να υπάρξει συνένεση για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγεία. Είναι σαφέ ότι η εθελούσια μέθοδο δεν έχει αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν να βρούμε μια σωστή λύση να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Μίλησαν όλοι οι συντονιστέ οι, οι αντικαταστάτε του. ΕΛΚ, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριο Κριστιαν Μπουζόε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, συγχαρητήρια για την πολύ καλή παρουσίασή σα. Υπάρχει όμω ένα θέμα με το οποίο δεν ασχοληθήκατε στην αναγκαστικά σύντομη εισαγωγή σα, που είναι πολύ μεγάλη, από τι μεγαλύτερε προκλήσει που έχουμε στα συστήματα υγεία μα. Είναι η ψηφιοποίηση. Δηλαδή υπάρχουν για παράδειγμα ηλεκτρονικές συνταγές, υπάρχουν ηλεκτρονικά ιστορικά, υπάρχουν τα κατάλληλα μητρώα, κυρίως για τον καρκίνο και την υπατήτητα, διαλειτουργικότητα, διαμεθοριακή ανταλλαγή στοιχείων, αλλά και χρήση της τηλεϊατρικής, της τεχνικής νοημοσύνης, της ρομποτικής. Πολλά πρέπει να κάνουμε σε πολλά κράτη-μέλη, αλλά και σε ενωσιακό επίπεδο η ψηφιακή υγεία εξελίσσεται ταχύτατα. Επαναλαμβάνω, βρίσκουμε νέες θεραπείες, αλλά κυρίως είναι θέμα καλύτερης οργάνωσης και πιο αποδοτικής χρήσης των πόρων στα συστήματα υγείας μας. Δηλαδή, η εξέλιξη των συστημάτων υγείας μας δεν μπορεί να γίνει χωρίς την καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Ως ε, μέλουσα ε, Επίτροπος Υγείας εάν σας εγκρίνει το Κοινοβούλιο, τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να ενισχύσετε την ψηφιοποίηση του κλάδου, του τομέα της υγείας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μποζούη για την ερώτησή σας. Όπως θα είδατε, στην επιστολή ανάληψης καθηκόντων, αναφέρομαι στην δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων. Η ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντικό τμήμα οποιοδήποτε θεματολογίου υγείας. είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτε μας. Είδαμε ήδη τα αποτελέσματα, γιατί ήδη πρόοδρος υπάρχει. Και θέλω να την χαιρετήσω. Για παράδειγμα, στην διαμεθοριακή υγεία, το 2019, για πρώτη φορά, βλέπουμε ηλεκτρονικές συνταγές μεταξύ δύο κρατών μελών. Και τα ιστορικά των ασθενών, επίσης, να είναι προσβάσιμα. Αυτό αποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρξει συνέχεια, πέρα από σύνορα της ε, θεραπείας αυτό το χρειάζονται οι ασθενείς. Δεσμευόμεθα να προωθήσουμε την ψηφιοποίηση ως Επιτροπή. Θα προτείνουμε έρευνα και ανάπτυξη από αυτού. Ήδη έχουμε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς, έτσι άτομα με σπάνιες ασθένειες και παιδικές ασθένειες έχουν τα στοιχεία τους προσβάσιμα. Αυτό μπορεί να αλλάξει ριζικά τη φροντίδα, τη θεραπεία των ασθενών. Βεβαίως δεσμευόμεθα πλήρω. Αλλά να προσθέσω και κάτι που ορισμένες φορές δεν αναφέρεται. Πρέπει να είμαστε επίση και προσεκτικοί, γιατί τίθενται θέματα προστασίας δεδομένων των ασθενών. Είναι κάτι που πάντα πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν θέτουμε το θέμα της ηλεκτρονικής υγείας. Η προστασία των δεδομένων είναι επίση σημαντική. ο Ευρωπαϊκός Χώρος ε, Στοιχείων Υγείας θα συνδυάσει όλα τα στοιχεία. Είναι τμήμα της επιστολής μου, της επιστολής ε, ανάθεσης καθηκόντων και θα συνεργαστώ με την ε, κυρία Φεστάγκερ για να το προωθήσουμε αυτό το θέμα τάχιστα. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται προστασία δεδομένων και για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Τίθεται και πολλά θέματα δεοντολογίας. Αλλά για να υπάρξει αυτή η διαλειτουργικότητα. Να υπάρχει ένα συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης των στοιχείων υγείας. Θα χρειαστούμε και την στήριξη των κρατών μελών και των πολιτών. Θα δώσετε περισσότερη πληροφόρηση στους ασθενούς για τα θέματα αυτά, για την ηλεκτρονική υγεία, για να έχουμε πιο αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη στο ίδιο σημείο, στο ίδιο επίπεδο. Για να προχωρήσουμε μαζί πρέπει να υπάρχει κάποια χρησιμότητα των επίπεδων. Δεν είναι από πλευρά ψηφιοποίηση όλοι στο ίδιο επίπεδο. Πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη, να βοηθήσουμε του βραδιπορούντε για να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν πρόκειται να εφαρμόσουμε την ε, διαμεθοριακή οδηγία που άλλαξε και βελτίωσε τη ζωή τόσο πολλών ασθενών. Γιατί πρέπει να δούμε και τι θετικό έγινε τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την ηλεκτρονική υγεία. Γνωρίζω τα προβλήματα και γνωρίζω και αυτό που αναφέρατε που δυστυχώς ε, αποσιωπείται πολλές φορές. Πρέπει να αυξήσουμε την πληροφόρηση προς τους ασθενείς. Πολλές φορές δεν γνωρίζουν ασθενείς τι δυνατότητες υπάρχουν για να τις αξιοποιήσουν. Είναι υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώνουν διαρκώς τους ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ. Από, τους ε, σοσιαλιστές, Ρόλι Πάντερ. Ευχαριστώ. Αν προωθήσετε ένα φιλόδοξο σχέδιο καρκίνου για την Ευρώπη, είμαι σίγουρος ότι το Κοινοβούλιο ενωμένο και αποφασισμένο θα σταθεί στο ύψος αυτό της ε, φιλοδοξίας για να δουλέψουμε μαζί. Σήμερα το βράδυ αναφέραμε συχνά την προ... τη σημασία της πρόληψης. Είναι σημαντισ... πολύ σημαντική για τον καρκίνο, αλλά και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία. Οποιαδήποτε προσπάθεια για ε, σχέδιο για τον καρκίνο ε, μπορεί να αντιβαίνει σε κάποια ισχυρά συμφέροντα του καπνού, ε, της παραγωγής χημικών, ε, υνοπνευματοδών ε, ποτών, ε, τη βιομηχανία των τροφίμων. Θα έχετε δύσκολες συζητήσεις που θα είναι απόσπαστο τμήμα αυτού του θεματολογίου. Τι στάση θα έχετε και τι μέτρα θα προωθήσετε για να μειώσετε την χρήση του καπνού και να υπάρχουν πιο ε, σωστά επίπεδα χρήσης του ινοπνεύματος στον πληθυσμό μας. Για το αν θα θελήσω να κάνω αυτή τη συζήτηση, βεβαίω. Θα θελήσω να χαμηλώσω τον πύχη σε αυτέ τι συζητήσει, όχι. Δεν πρέπει να χαμηλώσουμε τον πύχη όταν μιλάμε για την πρόληψη του καρκίνου. Ξέρουμε ότι μπορούμε να προλάβουμε πολλέ μορφέ καρκίνου που σκοτώνουν ανθρώπου. Θα πρέπει να δούμε το θέμα του καπνού. Υπάρχει ένα ε, κανονισμό για τον καπνό, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε έντονα. Έχει οδηγία για τον καπνό, διορθώνει η μιλήτρια, για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε επίπτωση και στους νέους, οι οποίοι δυστυχώς ε, όλο και περισσότερο στις μέρες μας χρησιμοποιούν καπνό και κινδυνεύει η υγεία τους. Επίσης, το ενόπνευμα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Οτιδήποτε υπάρχει στο περιβάλλον επηρεάζει την πρόληψη και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αν θέλουμε να δράσουμε σε επίπεδο πρόληψης. Το σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου είναι φιλόδοξο, αλλά πιστεύω ότι αν συνεργαστούμε μαζί με ευθύνη και υπευθυνότητα, μπορούμε να φέρουμε, να κάνουμε την αλλαγή. Σε καμία περίπτωση δεν θα διστάσω να επιτεθώ σε όσους δεν είναι υπέρ μιας προσπάθειας προ τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε. Ο καρκίνος αγγίζει την καθημερινότητά μας, την καθημερινότητα πολλών συμπολιτών μας. Και το είπα και στην αρχική μου παρέμβαση. Πρέπει να δούμε το θέμα σφαιρικά. Η πρόληψη είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της προσπάθειας και πρέπει να το δούμε και το θέμα και οριζόντια και να λάβουμε υπόψη μας και τον τρόπο ζωής. Γιατί ο τρόπος ζωής του καθενός είναι τμήμα της πρόληψης. Θα κάνω λοιπόν μεγάλη προσπάθεια στην ενημέρωση, στην ε, συνεργασία με τους ενδιαφέρομενους φορείς για την πρόληψη, για την αλλαγή του τρόπου ζωής, για να έχουμε πιο ασφαλή τρόφιμα. Ευχαριστώ. Εξορισμού η πρόληψη χρειάζεται χρόνο. Επανέρχομαι στο θέμα των θεραπείων καρκίνου. Εδώ και τώρα. Μπορείτε να πείτε λίγα περισσότερα για τις προσπάθειες που θα καταλάβετε για να υπάρχει ίση πρόσβαση σε θεραπείας καρκίνου σήμερα. Ε, με την προηγούμενη απάντηση σχεδόν δεσμευτήκατε να κάνετε ό,τι μπορείτε για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε απόλυτα το, το θέμα του πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Και Υπάρχει περίπτωση να αναθεωρήσετε τον κανονισμό για τα ορφανά και παιδιατρικά φάρμακα. Ο κανονισμός για τα παιδιατρικά και ορφανά φάρμακα αξιολογείται αυτή τη στιγμή. Είναι ένας κανονισμός που υιοθετήθηκε για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση των παιδιών και εκείνων με σπάνιες ασθένειες και για να έχουν περισσότερες θεραπευτικές επιλογές. Θέλω να δω το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις διασυνοριακές δοκιμές για τα παιδιατρικά φάρμακα και να δουλέψουμε όχι μόνο πάνω στο, στην αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, αλλά και πάνω στην ηλεκτρονική υγεία. Και τα ευρωπαϊκά δίκτυα υγείας κάνουν τη διαφορά. Νομίζω το 2016 υπήρξε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μίλαγε για τις ανισότητες θεωρώ ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις στρατηγικές μας εγώ προσωπικά. Θέλω να περιμένω όμως ε, για να δω λιγάκι. Νομίζω ότι πρέπει να βασίσω την προσπάθειά μου σε στοιχεία. Πρέπει να βγει πρώτα η αξιολόγηση του καονισμού, γιατί ο καονισμός αυτός έκανε τη διαφορά. Ευχαριστώ για το Renew Europe, ο Μάρτιν Χόζικ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας έχουμε εδώ, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, και χαίρομαι ιδιαίτερα και που το θέμα της πρόληψης του καρκίνου και της περιβαλλοντικής υγείας είναι υψηλά στις ε, γιατί πραγματικά είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό καθε αυτό, αλλά και η έλλειψη διαφάνειας και το πώ αντιμετωπίζουμε. Οι προλαλήσαντες ε, αναφέρθηκαν ε, στο πρόβλημα με τις μέλισσες ε, και την αδειοδότηση φυτοφαρμάκων. Και ακόμα και τους ενδοκρινικούς ρεταράκτες και όλα αυτά που ανέφερα, τα διέπει το ίδιο νήμα. Η έλλειψη διαφάνειας. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής σε μία ε, έκθεση στην Τεχνική Επιτροπή για τις Μεταφορές ε, ε, διαπίστωσε ότι υπήρχε παραβίαση διότι δεν υπήρχε πρόσβαση στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς προσωπικά για τις συστάσεις του Ευρωπαίου Μεσολαβητή προς αυτή την Επιτροπή και αν σκοπεύετε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία της επιτροπολογίας. Ευχαριστώ πολύ η διαφάνεια πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των όσων κάνουμε. Και αν ε, οι ομίγυροι είναι ειλικρινείς εδώ, ένας λόγος ε, για τον οποίο έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών ε, σε πολλά από αυτά που κάνουμε όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την καινοτομία και την προστασία έχει σχέση με το γεγονός ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει διαφάνεια σε πολλά από τα αποτελέσματα στα οποία θα έπρεπε ε, να έχουν πρόσβαση. Υπ' αυτή την έννοια ανέφερα και προηγουμένως ε, τις αλλαγές στη γενικότερη νομοθεσία για τα τρόφιμα ε, που βασίζονται στη διαφάνεια και ελπίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη σχέση εμπιστοσύνης ε, με τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Επίσης εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι πολλά από τα όσα συζητήσαμε προηγουμένως που έχουν σχέση με τις μέλισσες και το έγγραφο των κατευθυντηρίων γραμμών για τις μέλισσες δεν οφείλονται στην έλλειψη διαφάνειας αλλά στο γεγονός ότι τα κράτη-μέλη ε, αντιστέκονται και δεν τα εφαρμόζουν. Ε, και νομίζω ότι υπάρχουν και μια σειρά από πτυχές που πρέπει να εξετάσουμε και η διαφάνεια για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι χωρίς διαφάνεια δεν μπορούμε να έχουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και πολλά από αυτά τα οποία κάνετε εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο και πολλά από αυτά τα οποία ελπίζω ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα περάσουν εάν δεν υπάρξει αυτή η εμπιστοσύνη στις πολιτικές που προτείνουμε. Και ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του για αρκετούς λόγους ε, και στόχος μου είναι να προσπαθήσω να συνεργαστώ στενά με όλους τους ενδιαφερομένους προκειμένου να ανακτήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί. Ε, προσβλέπω πάρα πολύ στη συνεργασία μαζί σας. Πιστεύω σε αυτή τη συνεργασία. Μπορείτε να μας ε, δώσετε πολλά από αυτά που ε, ε, λένε οι πολίτες για να μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούμε καλύτερα σε αυτό που σκέφτονται. Ευχαριστώ. Ε, με ικανοποιεί ιδιαίτερα η δέσμευσή σας για τη διαφάνεια. Θα ήθελα λοιπόν ως επερώτηση να ρωτήσω εάν θα ζητήσετε κάτι τέτοιο από τα κράτη-μέλη, διότι πολύ συχνά οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται στις επιτροπές του Συμβουλίου ε, και κλεισμένων των θυρών. Θα ζητήσετε αυτές οι αποφάσεις να γίνονται αυτομάτως ε, δημόσιες και να μαθαίνουμε και πώς ψήφισαν τα κράτη-μέλη θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη προκειμένου να τους πείσουμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και θα προσπαθήσω να βρω και ε, λύσεις ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζω ότι έχουν υπάρξει προβλήματα, αλλά δεν είμαι αφελώς αισιόδοξη ότι με μια ειλικρινή συζήτηση θα καταφέρουμε να βρούμε τη σωστή λύση. Ε, η δουλειά μας δεν είναι να τιμωρούμε, η δουλειά μας είναι να βρούμε συνένεση και εγώ έτσι έχω μάθει να δουλεύω σε διάφορα επίπεδα και ευχαρίστως αναλαμβάνω αυτή την πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Από το ΕΛΚ τώρα, η Εύα Κόβατς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Κυριακίδου για τις ε, πολύ πλήρεις απαντήσεις του οράματός σας για τη δράση σας ως Επιτρόπου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Καρκίνου. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα το ότι έχετε ήδη απαντήσει πριν καν ε, τη θέσω. Οπότε να πω κάτι για την πολιτική για τα φάρμακα. Γιατί υπάρχουν λήψεις ε, πολλών αναγκαίων φαρμάκων, όχι μόνο αντικαρκυνικών. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν τα φθηνά φάρμακα. Οπότε, η ερώτησή μου είναι πώς θα λύσετε το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που είπα τόσα πολλά για το πρόγραμμα δράση για τον καρκίνο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό τμήμα της επιστολής που έλαβα. Για μένα είναι μια απίστευτη ευκαιρία να μπορέσω να εργαστώ εφόσον με εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων, έχετε δίκιο. Είναι τρομερό θέμα. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Αρχή Φαρμάκων έχουν κάνει μια ειδική ομάδα που ασχολείται με το θέμα αυτό. Θέλουμε να δούμε τι θα προκύψει από τις εργασίες της. Οι ελλείψει αυτές δεν, δεν οφείλονται σε ένα μόνο λόγο, αλλά σε πολλαπλού είναι θέμα τιμή, είναι θέμα επιστροφών εξόδων στους ασθενείς, είναι θέμα γενικότερα της φαρμακοβιομηχανίας. Θα έπρεπε να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης ε, προειδοποίησης για το που θα υπάρξουν ελλείψεις. Ένας λόγος που συχνά ακούω είναι ότι υπάρχει παράλληλο εμπόριο. Αυτό είναι ανησυχία. Αλλά δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε γενικά εντός της Ένωσης. Τα κράτη-μέλη, ωστόσο, θα μπορούσαν να περιορίσουν τις εξαγωγές αν υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων για κάποια φάρμακα στο εσωτερικό. Θα επιχειρήσω να το συνδυάσω με την πρόσβαση στα φάρμακα. Οι ελλείψεις και οι προσιτή τιμή είναι εξίσου σημαντικά θέματα. Για δύο λόγους. Πρώτον, ο φαρμακευτικός κλάδος έχει νομική υποχρέωση να επιτρέπει πρόσβαση των φαρμάκων στους ασθενείς, αλλά είναι και δικαίωμα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα σε προσιτή τιμή και ασφαλή. Δεν έχω τώρα μία έτοιμη απάντηση και λύση, αλλά ξέρω ότι πρέπει να δράσουμε σε διάφορα επίπεδα για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και κάτι πολύ σύντομα. Γίνεται τίποτα τώρα για την οικονομική συμβολή των φαρμακευτικών εταιριών προς, τον Ευρωπαϊκή, προς την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Φαρμάκων. Αν δεν γίνονται θα κάνετε κάτι γι' αυτό. Από ό,τι γνωρίζω, νομίζω ότι οι συζητήσεις αυτές είναι ανεξελίξη. Αλλά πρέπει να το ξαναδούμε, είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και θα ενεθάρρυνε και την καινοτομία, δηλαδή να προκύψουν νέα φάρμακα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ σοσιαλιστές και πράσινους και δημοκράτες, η Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ κύριε υποψήφια επίτροπε. Θέλω να επανέλθω στο θέμα των φυτοφαρμάκων. Είπατε ότι δουλεύετε βάσει επιστημονικών αποδείξεων. Υπάρχουν όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες που δείχνουν τη σχέση ανάμεσα στη χρήση των φυτοφαρμάκων και τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Αυτά τα φυτοφάρμακα τα καταπίνουμε, τα χρησιμοποιούμε ε, μέσω μολυσμένων φαρμάκων και νερού. Τα τελευταία χρόνια η πώληση φυτοφαρμάκων είναι σε σταθερά επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά δηλαδή τις μελέτες, οι χρήστες των φυτοφαρμάκων είναι πεπισμένοι ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένη από την απάντηση που δώσατε, γι' αυτό θα αναδιατυπώσω τις ερωτήσεις μου Πρώτον, πώς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι η οδηγία για τα φυτοφάρμακα μεταφέρεται σωστά στην εσωτερική νομοθεσία των κρατών μελών, γιατί είπατε ότι υπάρχουν προβλήματα εφαρμογή και ενσωμάτωση. Πώ θα εξασφαλίσετε ότι τα κράτη-μέλη κάνουν αυτό που πρέπει. Δεύτερον, πώ σκοπεύετε να μειώσετε την εξάρτηση που έχουν τα κράτη-μέλη στα φυτοφάρμακα. Μίλησατε πολύ για το σχέδιο δράση για τον καρκίνο. Μπορείτε να φτιάξετε και ένα σχέδιο δράση για να καταπολεμήσουμε τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Και πώς θα υποχρεώσετε τα κράτη-μέλη να περάσουν σε εναλλακτικέ λύσεις που υπάρχουν και που δεν βασίζονται στα χημικά. Θα θέσω τον, την ίδια ερώτηση τον κύριο Καμφάν για έναν στόχο με νούμερα για τη μείωση των φυτοφαρμάκων, γιατί πάνω σε αυτό δεν απαντήσατε. Και χωρίς αυτή την απάντηση δεν ε, μπορώ να πιστώ. Θέλω περισσότερες διευκρινήσεις απέναντι στην ερώτησή μου. Um, Θα επαναλάβω αυτό που είπα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να μ' ακούσετε. Είπα ότι δεσμεύομαι να μειώσουμε την εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα. Κάνω προσπάθεια γι' αυτό και να βρούμε νέες εναλλακτικές λύσεις με χαμηλότερο κίνδυνο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την επίπτωση που έχουν τα φυτοφάρμακα στην υγεία. Και θα ήταν πρωτάκουστο να είμαι επίτροπος υγείας και να μην ασχοληθώ με το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχει ισχυρή νομοθεσία στην Ευρώπη. Όμως δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Υπάρχουν συνεχείς έλεγχοι που γίνονται πρέπει να παρακολουθούμε τη δράση των κρατών μελών και να καταλάβουμε γιατί δεν εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία. Και όταν βλέπουμε ότι το πρόβλημα παραμένει, πρέπει να λάβουμε μέτρα. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω όμως είναι ότι αυτό δεν το βλέπω απομονωμένα από τα υπόλοιπα. Είναι τμήμα της Πράσινης Συμφωνίας που θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε όλοι και τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο. Το να το εντάξουμε αυτό το στοιχείο εκεί είναι σημαντικό για να έχουμε αποτελεσματική στρατηγική, πράσινη στρατηγική και στρατηγική από, το πιάτο στο, από την φάρμα στο πιάτο. Αν το δούμε απομονωμένα, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των φυτοφαρμάκων. Να συνεχίσω. Για τα χημικά προϊόντα, τα οποία είναι πολύ τοξικά, έχουμε νομοθεσία και χρησιμοποιούμε την επιτροπολογία για αυτά, ούτω ώστε συχνά ε, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα προϊόντα που είναι υψηλά τοξικά παρά τις μελέτες που υπάρχουν. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, τα χρησιμοποιούμε. Και μερικές φορές περνάνε και πέντε χρόνια. Αυτά τα χημικά, τοξικά προϊόντα παραμένουν στην ευρωπαϊκή αγορά για πάνω από πέντε χρόνια. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και δεν ενθαρρύνει και την βιομηχανία να βρει εναλλακτικά προϊόντα. Τι θα κάνετε για να ενθαρρύνετε τη βιομηχανία να βρει εναλλακτικά προϊόντα. Μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Να γίνει μια αξιολόγηση η οποία θα δείχνει την τοξικότητα αυτών των προϊόντων δηλαδή. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε στη γλυφοσάτη. Όχι μόνο. Κατάλαβα γιατί αυτή έλαβε έγκριση πενταετούς διάρκειας και είναι ε, μια ουσία η οποία μας διαιρεί πάρα πολύ και έχει ξεκινήσει τώρα η νέα αξιολόγηση. Χρειαζόμαστε διαφάνεια, πρέπει να βασίσουμε τις αποφάσεις μας σε επιστημονικά στοιχεία, θα συνεργαστώ για να υλοποιήσουμε τους στόχους της μείωσης και είναι πολύ σημαντική αυτή. Αυτά ως τμήμα της Πράσινης Συμφωνίας. Εγώ πιστεύω ότι είναι τμήμα της ε, ενιαίας αντίληψης για την υγεία. Επομένως, η απάντησή μου είναι ναι. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την καινοτομία, ούτως ώστε να χρησιμοποιούμε λιγότερο τοξικές ουσίες, ουσίες χαμηλότερου κινδύνου. Πρέπει να το εξασφαλίσουμε αυτό, ούτως ώστε οι αγρότες να μην χρησιμοποιούν χημικές ουσίες που είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Thank you. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, η Τίλη Μέτς. Κυρία υποψήφια επίτροπε, θα ήθελα να σας μιλή, ρωτήσω για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Η, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στεναρή άποψη επί του θέματος. Έχουμε κρίνει 36 αντιρρήσεις σε εγκρίσεις γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην προηγούμενη θητεία και όπως ξέρετε δεν υπήρχε ποτέ ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών υπέρ αδειών για γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να αποφασίσει και μέχρι τώρα η συνήθις απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτούς τους οργανισμούς είναι ναι. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να απαντά καταφατικά και υπάρχουν πάρα πολλοί αιτιολογημένοι ε, λόγοι για να ε, απαντήσουμε όχι. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να ακούσετε προσεπτικά τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα ε, αυτό. Ε, θα σταματήσετε να λέτε ναι στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς όταν δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία από αυτόν. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τους νέους γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι τον Ιούλιο του 2018 ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να χρησιμοποιούνται γενετικώ τροποποιημένοι οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω δεν έχει λάβει ακόμα μέτρα για να προστατεύσει του καταναλωτέ και του γεωργού από αυτά τα νέου γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Δεν θα πρέπει να περάσει αυτό το θέμα κατεπηγόντω και αξιολόγηση ασφάλεια, συχνηλασιμότητα και επισήμανση για αυτού του οργανισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι οι γενετικώ τροποποιημένοι οργανισμοί είναι ευαίσθητο και πολύ συχνά ένα θέμα που διχάζει. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ανεξάρτητα από αυτό που μας δείχνουν οι επιστημονικές ενδείξεις υπάρχει έλλειψη ε, των ε, ε των πολιτών για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Ε, εάν έχουμε βέβαια κατάλληλη εικόνα του τι ακριβώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε επιστημονικέ ενδείξει, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα. Οι αποφάσει πρέπει να βασίζονται στι επιστημονικέ ενδείξει. Ο ΕΦΣΑ, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό, δίνει έγκριση μόνο για ασφαλείς γενετικού τροποποιημένου οργανισμού, αλλά 19 κράτη-μέλη αποφάσισαν να περιορίσουν την καλλιέργεια γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών στην ε, χώρα τους. Επομένως, ε, δεν ε, λαμβάνουν υπόψη μόνο τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, αλλά και το τι αφορά τους πολίτες. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2018, τη σέβομαι απολύτως και πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή για τους οργανισμούς αυτούς που τροποποιούν το γονιδίωμα. Θα περιμένουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και να συνεργαστούμε μαζί σας και άλλους ενδιαφερομένους. Και σημείωσα ότι είπατε αν θα σεβαστείτε και θα πείτε ναι στη δημοκρατία και αν θα ακούσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην μπορώ να δεσμευθώ για πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεσμεύομαι για δύο πράγματα. Ναι, πάντα σέβομαι τη δημοκρατία και δεύτερον, και δεν είναι και κενά λόγια αυτά, θα ακούσω το Κοινοβούλιο και ε, ε, έχω την πρόθεση να είμαι διαθέσιμη και να συνεργαστώ στενά μαζί σας. Γιατί πολλά από αυτά τα θέματα, όπως οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί, όπως οι νέες τεχνολογίες ε, καλλιέργειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τόνισε και προώθησε ψηφίσματα τα οποία οδήγησαν σε αλλαγές. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τα κρατημέλη και τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους για να τα προωθήσω αυτά. Και πάλι, μπορεί να ακούγομαι μονότομη βέβαια, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι τμήμα της δικής μου στρατηγικής ε, το, από το χωράφι στο πιάτο. Συνεχίζω λοιπόν αμέσως. Είπατε ότι ε, εγκρίνουμε μόνο τους ασφαλείς γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού. ξέρουμε ότι υπάρχουν κενά στις αξιολογήσεις τη ΕΦΣΑ. Δεν εξετάζουν κατάλοιπα ε, φυτοφαρμάκους όπως ε, τη γλυφοσάτη που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή. Αλλά απαντήσατε στην ερώτηση για την δημοκρατική νομοποίηση και χαίρομαι γι' αυτό. Όσον αφορά την λασιμότητα όμως των νέων γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μεθόδους ανείχνευσης το συντομότερο δυνατόν και πρέπει εσείς να ανοίξετε το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Δεσμεύεστε να κάνετε κάτι τέτοιο. Καταρχάς γνωρίζω ότι η ΕΦΣΑ είναι υπό την αρμοδιότητά μου, την πολιτική και δεν θα διστάσω αν διαπιστώσω ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσω, να το εξετάσω. Το δεύτερο είναι ότι εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω τις νέες τεχνικές ε, αναπαραγωγής ε, για τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουμε ε, και τις ενδείξεις που θα έχουμε και αν πρέπει να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο, σαφώς χωρίς δισταγμό θα το εξετάσω. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν μας εμπιστεύονται, αλλά γνωρίζω ακόμα περισσότερο ότι οι πολίτες ανησυχούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει διαφάνεια, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν αυτό που τους προσφέρουμε. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν από πού προέρχεται τα τρόφιμα στο τραπέζι τους και σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Λαντσίνη, από ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανησυχία για τις απάτες στα τρόφιμα και την ε, ε, ποιότητα των τροφίμων υποσκάπτουν την υγεία και την εμπιστοσύνη των, ε, καταναλωτών. Δημιουργούν πρόβλημα από τους γεωργούς, εμπιστοσύνη απέναντι στους γεωργούς. έχουμε διάφορες απάτες το 2017. την απάτη στο Βέλγιο που πουλούσαν κρέας αλόγου για, αντί για κρέας βόηου. 100 ε, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ε, μας κοστίζουν αυτές οι απάτες. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν πολύ περισσότερο, λειτουργούν στα πιο αδύναμα κράτη-μέλη που δεν έχουν καλούς ελέγχους. Οι ποινικέ κυρώσεις δεν είναι επαρκείς για να λύσουν αυτό τα προβλήματα και δεν υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις. Υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων στη Γενική Διεθνήση Άγκρη και Σάντε και υπάρχει ε, ο κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους του 2017, άρθρο 108, όπου η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τους κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών. Πώς προτίθεται η Κομισιόν να βελτιώσει το σύστημα πρόληψης και εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Thank you, thank you for that question. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Η απάτη στα τρόφιμα κοστίζει 8 με 12 δισεκατομμύρια. Επηρεάζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Δυστυχώς από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει νομικός ορισμός της απάτης στα τρόφιμα. Είναι απάτη, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το 2013, αν την ένα ψήφισμα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη Europol, το Γραφείο Καταπολέμησης των Απατών, για να εντοπίσουμε τις απάτες αυτές και βεβαίως επιθυμώ να συνεργαστώ με όλους για να δούμε μήπως θέλουμε νέα νομοθεσία για να ελέγχουμε το πρόβλημα. Μικρόφωνο. Ο λόγος για τον οποίο η ασφάλεια των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να αξιολογείται είναι γιατί χημικές ουσίες μπορεί να περάσουν στα τρόφιμα και να υποσκάψουν την υγεία των καταναλωτών. Η σχετική νομοθεσία, ο κανονισμός 1935 του 2004, είναι μια καλή νομική βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αφορά λίγα, λίγες ουσίες όπως τα πλαστικά. Μόνο εκεί υπάρχουν εναρμονισμένα μέτρα. Πολλέ ουσίε ρυθμίζονται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Αυτό δημιουργεί μια ανομοιομορφία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Και βεβαίω και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η Κομισιόν τους, ε, τα επόμενα χρόνια προτίθεται να υιοθετήσει εναρμονισμένα μέτρα και για άλλε ουσίε πέραν των πλαστικών. Ε, Ευχαριστώ. Ε, σε, αναφέρεστε σε ουσίες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτές οι ουσίες μπαίνουν στα τρόφιμα και πιθανώ επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία αλλά και, τη σύνθεση, και αλλάζουν και τη σύνθεση των τροφίμων. Υπάρχει ένας κανονισμός του 2004 για αυτό το θέμα που αξιολογείται αυτή τη στιγμή και γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο το 2016 ζήτησε να αξιολογηθούν άλλες 13 ουσίες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πιθανώ. Οι κανόνες που ακολουθούν, τα κράτη-μέλη διαφέρουν, ισχύει αυτό. Έχουμε πληροφορίες από εκθέσεις που δημοσιεύονται για τα πλαστικά, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες για πολλέ άλλε ουσίες. Θέλω να προσθέσω και κάτι. Η ΕΦΣΑ εξετάζει αυτό το θέμα, αλλά να σας πω και κάτι επιπλέον θα πρέπει να έχουμε πληροφορίες για την επίπτωση που έχουν τα κοκτέιλ αυτών των ουσιών όταν έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει επίσης πολύ σημαντικά την υγεία. Αν σκοπεύουμε να νομοθετήσουμε, όπω ρωτήσατε, και άλλε ουσίες, καταλαβαίνω την ανησυχία, θα κοιτάξω τι επιστημονικά στοιχεία έχουμε, θα κάνουμε μια ιεράρχηση των στόχων μας, θα ξεκινήσουμε από τις ουσίες που είναι πιο επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Είναι πάντως ένας πολύ σημαντικός τομέας. Εντάσσεται όχι μόνο στρατηγική για, από το χωράφι στο πιάτο, αλλά και την Πράσινη Συμφωνία. Έρμαν Τέρτσο από την ομάδα συντηρητικών και, μετα... και μεταρρυθμιστών. Καλησπέρα σας κυρία Κυριακίδου. Ζούμε σε δύσκολου καιρού. Η επιστήμη και η τεχνολογία πολλέ φορέ περιθωροποιούνται γιατί η συζήτηση γίνεται με συναισθηματικού όρου και πολλή παραπληροφόρηση. Και δεν λαμβάνουν ε, οι, αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις επαρκώς την επιστήμη υπόψη. Ο κύριος Ανδριοκάητης ε, ήταν ε, από τους λίγους που υπερασπίζονταν την επιστήμη. Ούτε ο πρώτος Γιούνκερ, ούτε οι άλλοι επίτροποι τον στήριξαν στην σταυροφορία του κατά του φανατισμού που είναι κατά της επιστήμης. Πώς θα κερδίσετε λοιπόν την υποστήριξη των άλλων επιτρόπων, γιατί είναι πολύ δυσχερές το έργο σας να στηρίξουμε τα επιστημονικά δεδομένα, στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως. Τελικά, κυρία υποψήφια επίτροπε, ποιες είναι οι συγκεκριμένε αντιλήψεις σας, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το ρόλο που παίζει η επιστήμη έναντι στην πολιτική και τις ιδεολογικές προκαταλήψεις στην νομοθετική διαδικασία. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι οι αποφάσεις πολιτικής πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη. Αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Δεν το αποδέχονται ορισμένες φορές οι πολίτες λόγω του επίπεδου παραπληροφόρησης. Παράδειγμα, έχουμε τα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι πρέπει να εμβολιαζόμεθα όμως τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε μια σειρά από ασθένειες να επανέρχονται στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα η λαρά, λόγω αυτής απροθυμίας εμβολιασμού. Δεν θα πω ότι αυτό οφείλεται μόνο σε παραπροφόρηση. γιατί έχει να κάνει και με τα προγράμματα των κρατών μελών για τον εμβολιασμό. Δεν υπάρχει ομοιογένεια σε αυτά. Αλλά υπάρχει τώρα κοινή δράση της Ένωσης γι' αυτό και μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον έλεγχο και την πρόληψη των ασθενών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Φαρμάκων πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε πηγή παραπληροφόρησης που έχει επίπτωση τελικά, αρνητική βέβαια, σε περιπτώσεις που έχουμε επαρκή επιστημονικά στοιχεία. Ο στόχος μου θα ήταν να, είμαστε μια να είμαι μια υπεύθυνη φωνή στο σώμα των επιτρόπων, η επιστήμη, τα στοιχεία να είναι η βάση των αποφάσεών μας, λαμβάνοντας υπόψη και αντιμετωπίζοντας και άλλες ανησυχίες για να μπορέσουμε να πείσουμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται πολλές πολιτικές που ξέρουμε ότι είναι αναγκαίες για να προστατεύσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια. Ορισμένοι δεν περιμέναμε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δυστυχώ λοιπόν τα τελευταία χρόνια η παραπληροφόρηση μα έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για να προωθήσουμε θέματα που έχουμε επιστημονικά στοιχεία. Αυτή η παραπληροφόρηση όμω έχει και άλλα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι. Οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, όπω είναι και η έρευνα, χρειάζεται μακροπρόθεσμη πολιτική, ασφάλεια. Η έρευνα και ανάπτυξή μας στον ε, αγροεπιστηστικό τομέα, για παράδειγμα, εγκαταλείπει την ε, Ένωση. Έχουμε διαρροή εγκεφάλων ε, όλο και πιο έντονη. Αυτό οφείλεται στην ομοθεσία που πολλές φορές δεν βασίζεται στην επιστήμη. Και πολλές φορές αυτή η αρχή της προφύλαξης χρησιμοποιείται υπερβολικά για λόγους ιδεολογικοπολιτικούς. Νομίζω ότι κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Θεωρούμε ότι τα φυτοφάρμακα, για παράδειγμα, είναι ο διάβολος, ενώ για ορισμένα θέματα δεν έχουμε εναλλακτικέ λύσει. Έτσι, δεν αναπτύσσουμε και νέε στρατηγικές της τροποποίηση του γονιδιώματο, για παράδειγμα. Προτίθεστε να επανεξετάσετε την αρχή της προφύλαξη. Και είστε τεθειμένοι να υπερασπιστείτε την καινοτομία που την χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι παγκόσμιος ηγέτη στα θέματα αυτά. Μα είναι απόλυτη υποχρέωσή μας να είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες. Η Ευρώπη πρέπει να ηγείται σε πολλούς τομείς που σχετίζονται με την υγεία και για την ε, επιστημονική έρευνα και την καινοτομία, σίγουρα. Γνωρίζω ότι στο παρελθόν Λόγω τη οδηγία για τι κλινικέ δοκιμέ, τώρα δεν θυμάμαι ποιο χρόνο ενεκρίθη, είχαμε πολλέ δυσχέρειε για να οργανώνονται κλινικέ δοκιμέ. Οπότε οι περισσότερε τέτοιε δοκιμέ και μελέτε γίνονταν στι ΗΠΑ και αρχίσαμε να καθυστερούμε στην έρευνα. Αλλά αλλάξαμε την οδηγία. Τώρα μπορούμε να έχουμε περισσότερες κλινικές μελέτες στην Ευρώπη. Δεσμευόμεθα να προωθήσουμε την καινοτομία. Και δεσμευόμεθα για περισσότερες επενδύσεις. Το πρόγραμμα Horizon 2020 ήδη είναι η απόδειξη αυτής της δέσμευσης. Σίγουρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι προτεραιότητά μας αυτό, διότι η καινοτομία με βάση την επιστήμη θα έχουν θετικά αποτελέσματα για την υγεία στην Ευρώπη. Θα βοηθήσει τον κλάδο, θα μας επιτρέψει να βρούμε νέα φάρμακα, θα βοηθήσει την επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας, θα βελτιώσει τα τρόφιμά μας. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει και να παραμείνει ηγέτης και στην φαρμακοβιομηχανία. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως η ελλείψη φαρμάκων και ε, να έχουμε φάρμακα σε προστή τιμή. Δεσμευόμεθα σε αυτά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας ή ε, δυνατόν. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Αρλούκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι μπροστά σας, στο κέντρο, στην πρώτη σειρά. Στη διάρκεια αυτής της θητείας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και για σας ε, ως ε, Επίτροπο, μας αφορά όλους μία τεράστια πρόκληση. Κατά πόσον θα βρούμε το σθένος να αντιμετωπίσουμε τον πραγματικό δολοφόνο των Ευρωπαίων, τον καρκίνο. Εγώ είμαι γιατρός και για πάρα πολλά χρόνια ασχολήθηκα ε, με παιδιατρική ογκολογία. Και ως πρώην Υπουργός Υγείας γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αν τα κράτη-μέλη μείνουν μόνα τους, μόνο με τους πόρους που διαθέτουν για να καταπολεμήσουν τον καρκίνο, ποτέ δεν θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Υπάρχουν προδιαγραφές και πρωτόκολλα για ογκολογικές ε, θεραπείες για τα παιδιά, αλλά δεν υπάρχουν αντίστοιχες προδιαγραφές και πρότυπα για τους ενήλικες. Εάν λοιπόν ε, δεν αναλάβουμε αυτή την πρόκληση, οι άνθρωποι δεν θα μας ε, συγχωρήσουν ποτέ. Θα πρέπει να υπάρχουν πρότυπα για έγκαιρη διάγνωση και σύγχρονους τρόπους ε, θεραπείας ε, των ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Αυτές είναι οι προκλήσεις που έχουμε να εντοπίσουμε από κοινού και εσείς και εμείς και αυτό φυσικά είναι καθήκον ζωής. Ευχαριστώ. Κύριε Αρλούκοβιτς, δεν θα προσπαθήσω καν να μπω στη θέση κάποιου που προσπαθεί να πει ότι δεν έχει τα απόλυτο δίκιο, αλλά ε, θα ήθελα να προσθέσω και το εξή. Υπάρχουν πρωτόκολλα για τη θεραπεία για τους ασθενείς ε, που πάσχουν από καρκίνο, αλλά δεν ε, τα ακολουθούμε πάντα αυτά τα πρωτόκολλα και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ακολουθούμε τα πρωτόκολλα. Και όταν αναφερόμαστε σε σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, πρέπει να δούμε όλο το φάσμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, ξέρουμε ότι ε, οι διαγνωστικές εξετάσεις σώζουν ζωής. Ε, η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές, αλλά δεν αρκεί απλώς η διαγνωστική εξέταση. Πρέπει να υπάρχουν και διαγνωστικά προγράμματα τα οποία θα είναι επιστοποιημένα και που θα τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αυτό το οποίο εξέδωσε ψήφισμα που ορίζει τι θα πρέπει να καλύπτουν και ποια κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται από τα προγράμματα διάγνωσης. Ε, και πρέπει εμείς να φροντίσουμε να εφαρμόζονται αυτά. Συμφωνώ πολύ τους μαζί σας. Ο καρκίνος είναι για πολλούς μία νόσος που επηρεάζει όχι μόνο τον ασθενή αλλά και την οικογένεια, τον εργοδότη Υπάρχουν θέματα που κανένας ε, δεν αναφέρει. Η επιβίωση από τον καρκίνο. Τι γίνεται με χιλιάδες ασθενείς ε, μετά από τον καρκίνο. Πώς τους αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους. Ε, τι ασφάλεια υγείας δικαιούνται εάν πούνε ότι έχουν υπάρξει ασθενείς καρκίνου. Είναι τεράστιο το φάσμα. Γι' αυτό και ακριβώς η πρόκληση είναι να υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, το οποίο αναφέρεται ρητός ε, στην επιστολή της αποστολή μου. Ε, το Κοινοβούλιο έχει κάνει πάρα πολλά. Υπάρχει Επιτροπή των Μελών κατά του Καρκίνου. Έγινε εξαιρετική δουλειά και προωθήσαμε πάρα πολλά πράγματα και τώρα μπορούμε να τα προωθήσουμε έτσι περαιτέρω. Στην ε, Πολωνία εγώ ήμουν αυτός ο οποίος εισήγαγε την ε, περιβόητη δέσμη μέτρων ε, για τον καρκίνο ε, που σημαίνει ότι ελήφθησαν αποφάσεις για χρηματοδότηση από το δημόσιο κορφανά για όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνουν γιατροί και κλινικές που ακολουθούν τα πρωτόκολλα και παρέχουν έγκαιρη διάγνωση. Και φυσικά δεν υπήρχε κανένας περιορισμός όσον αφορά τις δαπάνες και τα κονδύλια που τους δώσαμε. Αλλά το 2007 πολλά ε, κρατη το 2012 συγγνώμη, πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίσαν ελλείψεις σε φάρμακα για τον καρκίνο και ε, κινδύνεψαν να χαθούν ανθρώπινα ζωές. Ε. Θα λάβετε μέτρα για να μην υπάρχουν έλλειψη φαρμάκων και να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο γιατί στις ογκολογικές θεραπείες ο χρόνος είναι ε, ε κρίσιμος. Ευχαριστώ πολύ. Είχα και την χαρά να επισκεφθώ τη χώρα σας και να συνεργαστώ στενά με ιατρούς ε, και άλλους για να δούμε τα προγράμματα διάγνωσης τα οποία εφαρμόζονται και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι ε, άνοιξαν και το δρόμο για πολλές άλλες χώρες το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την ε, ε, Καταπολέμηση του Καρκίνου ε, χρειάζεται ένα ολόκληρο φάσμα θεμάτων. Κάποιος συνάδελφός σας μίλησε για την πρόληψη, αναφέρομαστε στην πιστοποίηση και στα πρότυπα και αυτό φυσικά θα πρέπει να περιλαμβάνει και φάρμακα. Και γνωρίζω ότι πάρα πολλά κράτη-μέλη έχουν αντιμετωπίσει δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν και σε προβλήματα στην υγεία. Ε, ο κλάδος ε, των φαρμάκων και ο τομέας της υγείας θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα είναι προσιτά τα φάρμακα και φυσικά αυτό θα είναι στα σχέδιά μου και θα γίνουν κάποια πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να μειώσουμε, να κατεβάσουμε τον πύχη ε, με κανένα τρόπο σε αυτές τις αποφάσεις. Ευχαριστώ για το Renew η Caroline Βόντεν. Κυρία Κυριακίδου, εδώ είμαι. Το άρθρο 168 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία λέει ότι θα αναλάβουμε δράση για να προλάβουμε την, τις επιπτώσεις στην φυσική και πνευματική υγεία. Επί 20 χρόνια ήσασταν κλινική ψυχολόγος. Ένας στους έξι ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν πρόβλημα ψυχικής υγείας το 2016 και όλα τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι η ψυχική υγεία επηρεάζουν δεκάδες χιλιάδων Ευρωπαίων κάθε χρόνο. Υπάρχει πρόβλημα στι οικογένειε του και με την παραγωγικότητα. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, υπάρχει μια επιδημία προβλημάτων διαταραχής σε παιδιά και ενήλικες, κατάθλιψη, ε, διατροφικές διαταραχές, ε, τάση για αυτοκτονία. Τι θα κάνετε για να βάλετε την ψυχική υγεία ξανά στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο και τι συγκεκριμένα βήματα θα πάρετε, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις πολιτικές για την ψυχική υγεία και τις συστάσεις που υπάρχουν για την ψυχική υγεία. Προηγουμένως, όταν απάντησα σε κάποιες ερωτήσεις για άλλα θέματα, είχα πει ότι υπάρχει νέα αντίληψη για την υγεία. Την ε, υγεία των ζώων, την ε, ανθρώπινη υγεία και την υγεία των φυτών. Όταν μιλάμε για την ανθρώπινη υγεία, δεν μιλάω μόνο για το σώμα, τη σωματική υγεία, αλλά και την ψυχική υγεία γιατί είναι αλληλένδετα. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η ψυχική υγεία δεν είχε μπει στο θεματολόγιο για πολλά χρόνια, για πολλούς λόγους. Σε πολλά κράτη-μέλη στιγματίζονται οι ασθενείς. Ο κόσμος δεν αναζητάει βοήθεια αρκετά νωρίς. Αλλάζουν επίσης και οι πιέσεις απέναντι στα παιδιά και στους εφήβους. Βομβαρδίζονται από πληροφορίες που ο βαθμός ορίμανσής τους δεν τους επιτρέπει να φιλτράρουν σωστά κατά ανάγκη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτω ώστε να ξαναμπεί αυτό το θέμα στην ατζέντα μας. Γιατί πιστεύω ότι η ψυχική υγεία είναι ένα τομέα που για πολλά κράτη-μέλη Παραβλέπετε, Είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι για να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Και δεν μιλάω μόνο για την κατάθλιψη σε ενήλικους εδώ. Α, κοιτάξτε τα προβλήματα που έχουν οι έφηβοι. Προβλήματα συμπεριφοράς. Όλο και περισσότερο αυτοκαταστροφικές τάσεις και συμπεριφορές. Πρέπει να δράσουμε προληπτικά. Θα πρέπει όχι μόνο να λάβουμε υπόψη την υγεία τους, αλλά να δράσουμε και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Ε, πάνε στο σχολείο. Θα πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημά τους πολύ νωρίς, ούτω ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις, τη μελλοντική μου προσπάθεια και το χαρτοφυλακιό μου. Με ενδιαφέρον άκουσα να λέτε ότι είναι σημαντικό για σας, αλλά επί δύο ώρες πρώτη φορά ακούγεται ο όρος ψυχική υγεία και κανένας άλλος δεν το ανέφερε και μου κάνει εντύπωση αυτό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, ε, ορισμένοι είναι περιβαλλοντικοί, άλλοι είναι τα φάρμακα. Εσείς πώς θα συνεργαστείτε με άλλους επιτρόπους για να εξασφαλίσετε ότι η πίεση στο σχολείο, οι σεξουαλικές επιθέσεις, κακές σύνδικες εργασία, ε, κακή στέγαση, απομόνωση, όλα αυτά τα στοιχεία θα βελτιωθούν, ούτω ώστε να έχουμε λιγότερε περιπτώσει ψυχική υγεία στην Ευρώπη. Λέτε ότι θα κάνετε το καταδύναμη. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα, θέλω να, να μου πείτε. Θα έχετε, επενδύσετε χρήματα, θα υπάρξουν προγράμματα, θα γίνει κατάρτιση σε κράτη-μέλη και εκπαίδευση κρατών μελών που το θέμα της ψυχικής υγείας δεν είναι ψηλά στην ατζέντα τους. Τι θα κάνετε. Η συνεργασία με τους άλλους επιτρόπους είναι πολύ σημαντική, γιατί η ψυχική υγεία αφορά πολλούς τομείς όπως αναφέρατε κι εσείς. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν έχει ενδεχομένως την ευκαιρία να εξετάσει ποια είναι αυτά τα προβλήματα και τι πρέπει να αλλάξει. Είπατε ότι κανένα άλλο ε, δεν ανέφερε προηγουμένω ε, την ψυχική υγεία. Εγώ την ανέφερα στην αρχική μου παρέμβαση, γιατί τη θεωρώ σημαντική. Και την ανέφερα, γιατί πιστεύω ότι ένας από τους ε, λόγους που δεν γίνονται τόσα πολλά σε αυτό τον τομέα είναι ότι ξεχνάμε λιγάκι, βάζουμε στο περιθώριο αυτά τα άτομα. Πολλά πράγματα επηρεάζουν την ψυχική υγεία, συμφωνώ. Θα συνεργαστώ με άλλους ε, επιτρόπους, ούτω ώστε το θέμα της ε, ψυχικής υγείας να ενταχθεί σε πολλές πολιτικές. Και ελπίζω να μιλήσω για αυτό το θέμα και να εκπροσωπήσω όλους όσους πάσχουν από αυτό. Ευχαριστώ. Μη γεγραμμένη. Ο κύριος Κωνσταντίνου. Μιας και ο λόγο περί διανοητικής υγείας, από την προλαλήσασα, θα επιθυμούσα να καταθέσω από ιατρική σκοπιά μια πολυδύναμη ερώτηση σχετικά με την επικειμένη ενδεχομένη παρέμβασή σα ως Επιτρόπου Υγείας. Θα επιτρέψετε και θα υποστηρίξετε την εκπαίδευση και την έρευνα στην ιατρική και ειδικότερα στην ψυχιατρική σχετικά με τα ακόλουθα θεμελιώδη ζητήματα επιρροή ενός εκάστου εθνικού πολιτισμού επί του τι θεωρεί μια κοινωνία ω φυσιολογικό, παθολογικό ή ανώμαλο. Πιστοποίηση τη παγκοσμιότητα των νοσολογικών κριτηρίων και κατηγοριών τη βιοιατρική και της ψυχιατρικής σε διαφορετικού εθνικού πολιτισμού. Ταυτοποίηση και περιγραφή νοσημάτων που ανήκουν σε ειδικού πολιτισμού, γνωστών ω εθνικέ διαταραχέ ή ω συνδεόμενα προ τον πολιτισμό σύνδρομα όπω για παράδειγμα η νευρική ανορεξία ή το προεμινοπαυσιακό σύνδρομο στι δυτικέ κοινωνίε. Συσχετική επιρροή γονοτυπικών και φαινοτυπικών παραγόντων επί της προσωπικότητας και επί συγκεκριμένων μορφών ψυχιατρικών και ψυχοσωματικών παθολογιών. Τελειώνοντας, οφείλω να υπενθυμίσω ότι τα αναφερθέντα δεν αποτελούν αστήρικτες αναζητήσεις, αλλά υποστηρίζονται πολλοί από τη διεθνώς χρησιμοποιούμενη πέμπτη έκδοση του DSM του 2013, όπου συμπεριλαμβάνεται η συνέντευξη πολιτιστικής σχηματοποίησεως για την συγκεκριμενοποίηση της διαγνωστικής προσέγγισης των κλινικών συναδέρφων. Επίσης, ανάλογο βαρύνουσα σημασία mm-hmm. έχει το σχετικό πρωτοποριακό πόνημα των κ. Μάγκερ και Ρουσό πολιτιστική συμβουλευτική αντιμετώπιση. Sorry, Mr. President. Five seconds. Can I have it? Five seconds. Yes, just to fulfill the title. It's enough Ολοκληρώσω τον τίτλο. Και αντιμετώπιση αντιμετωπίζοντα τον άλλο στη φροντίδα θεματική υγεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. I don't dare say I didn't... Δεν μπορώ να πω, δεν τολμώ να πω ότι δεν την κατάλαβα, αλλά θα προσπαθήσω να την αντιμετωπίσω όσο προσεκτικά γίνεται. Ξέρω ότι το DSM έχει αλλάξει την ταξινόμηση των ψυχιατρικών ή άλλων προβλημάτων. Ξέρουμε ότι διάφορες διαταραχές που δεν θεωρούνται ψυχιατρικές, συγγνώμη, μάλλον που θεωρούνται τώρα έχουν εξαιρεθεί. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζουμε αυτό και πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς οι διάφορες κοινωνίες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα. Αναφερθήκατε στην ανορεξία. Δεν αναγνωρίζεται από άλλες, ορισμένες κοινωνίες. Και άλλες την αναγνωρίζουν και θεωρούν ότι έχει μεγάλες διαστάσεις. Βάση της προσέγγισής μου θα ήταν ότι πρωταρχικό για μένα είναι η προστασία και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι στην ψυχιατρική αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα λεπτό γιατί είναι πολύ εύκολο να βάλεις ταμπέλες στους ανθρώπους, να τους κολλήσεις μια ψυχιατρική διάγνωση. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ υποκειμενικό, ανάλογα με τον πολιτισμό της κοινωνίας όπου ζει ο κάθε ασθενής. Θα το εξετάσω πολύ προσεκτικά. Το τι είναι φυσιολογικό. Αναφερθήκατε στο τι είναι φυσιολογικό. Και αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί ορισμοί για το ότι είναι φυσιολογικό. Και θα χρειαζόμουν πολύ παραπάνω από δύο λεπτά για να το συζητήσω. Αλλά ευχαρίστω να το συζητήσω κάποια άλλη στιγμή μαζί σας. Ευχαριστώ κυρία Κυριακίδου. Απαντήσατε στην ουσία της ερώτησης. Ωραία συμπροματική. Για τους σοσιαλιστές. Η Σάρα Σέρντας. Κύριε υποψήφια επίτροπε, η ερώτησή μου ε, έχει να κάνει με 33.000 θανάτου και μας κοστίζει 1,1 η αντιμικροβιακή εντοχή συγκεκριμένα λοιπόν. Αυτό έχει να κάνει και με την κατάχρηση αντιβιωτικών χωρίς ε, συνταγές ή χωρίς να σέβονται οι ασθενείς την σύμβολη, την συμβουλές των ιατρών. Επίσης είπατε ότι επανέρχονται ασθένειες που τις είχαμε ξεπεράσει λόγω μείωσης της, ε, το, του εμβολιασμού. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν καλύτερα οι συμπολίτε μα ε, ποια είναι τα θέματα αυτά για να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση κατά των εμβολιασμών και να ε, διασφαλίσουμε ότι οι συμπολίτε μας χρησιμοποιούν σωστά την πληροφόρηση. Τι θα κάνετε για να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και σωστότερη χρήση των πληροφοριών. Θίξατε δύο θέματα που συνδέονται άμεσα. Έτσι έχουν να κάνουν τι σημαίνει γνώση, σωστή χρήση της ιατρικής προφόρησης και παραπληροφόρηση. Δυστυχώς, ένα από τα λατώματα της ψηφιακής εποχής είναι πόσο εύκολο είναι να διαδοθεί η παραπληροφόρηση. Υπάρχουν ε, τόσο πολλές δυνατότητες, τόσο πολλά κανάλια. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε πολύ στενά με τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες έχουν αξιόπιστη επιστημονική πληροφόρηση και όπου υπάρχει παραπληροφόρηση να την εντοπίζουμε τάχιστα. Αναφερθήκατε στην ε, αντίσταση στα αντιβιωτικά. Αυτό είναι τρομερό και παγκόσμιο πρόβλημα. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο ηγέτης μέσω της πρακτικής της στην αντιμετώπιση του, του θέματος αυτού. Είναι στο θεματολόγιο για την ενιαία προσέγγιση για την υγεία τη μία υγεία όπως λέμε, δεν είναι δυνατόν να πεθαίνουν 33.000 άτομα το χρόνο στην Ένωση για αυτό το λόγο. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να πεθαίνουν παιδιά από ασθένειε πριν από μερικά χρόνια τις είχαμε κρυζώσει στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε μέσω της εκπαίδευσης και μέσω των συστημάτων υγείας για να διαψεύσουμε την παραπληροφόρηση που όντω διαδίδεται και που έχει ουσιώδη επίπτωση στην υγεία των συμπολιτών μας. Ναι. Η φυματίωση. Τα θύματα της φυματίωσης ε, έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με την ε, αντίσταση στα μικρόβια και πολλοί από τους ασθενείς ε, φυματίωσης αναπτύσσουν αντίσταση σε πολλά φάρμακα και πεθαίνουν. Και επίσης ε, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έκλεισε την ειδική ομάδα μελέτης για το AIDS και για, έκλεισε επίσης το φόρουμ για το HIV, τη φυματίωση και την υπατήτηδα. Τι θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα δημόσιας υγείας αν δεν έχουμε αυτούς ε, τους ε, πολύ σημαντικούς συμπληρογνώμενους αυτών των δύο φορέων. Πιστεύω ότι υπήρξε ένα θαυμάσιο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το HIV, την υπατήτηδα και τη φυματίωση το 2017. Και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για αυτό το ψήφισμα, γιατί αυτές οι τρεις ασθένειες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς και μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά και για να τις προλαμβάνουμε. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την, τον έλεγχο και την πρόληψη των ασθενειών βοηθά τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες αυτές. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση στην καινοτομία και στα κατάλληλα φάρμακα για τους ασθενείς αυτών των τριών ασθενειών. Και υπενθυμίζω, το G7 στη συνάντηση του Biarritz δεσμεύτηκε να δαπανηθούν 550 εκατομμύρια για την καταπολέμηση αυτών των τριών ασθενών. Θα τους πιέσω να τα διαθέσουν, γιατί θίγουν πολλούς συμπολίτε μας αυτές οι ασθένειες. Αυτό θα ήταν η κύρια προτεραιότητά μου. Ευχαριστώ πολύ. Για το ΕΛΚ, ο Ντάνιελ Μπούντα, από την Επιτροπή Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, εγώ είμαι από την Επιτροπή Γεωργίας και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια τώρα για την υγεία των ζώων, η οποία για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και αυτό φυσικά έχει και τεράστιο αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και πιστεύω ότι και εσείς θα πρέπει να ασχοληθείτε με τα θέματα αυτά. Ο... Αυτό δυσπυρετός είναι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη ε, και η πανόλη των χείρων επίση, και δεν έχει γίνει κάτι για να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη νόσο. Πρόσφατα ε, είχαμε μεγάλη αύξηση στον αριθμό των περιστατικών. Φέτος ε, είχαμε μόνο 1.470 νέα περιστατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ελοχεύει ο κίνδυνο, το συντομότερο δυνατόν ο ιός αυτός να επεκταθεί και στη Δυτική Ευρώπη. Υπάρχει ανησυχία λοιπόν μεταξύ των κτηνοτρόφων και των εμπειρογνωμόνων σε θέματα υγείας των ζώων για τον αντίκτυπο που θα υπάρχει για τον κλάδο. Και πρόκειται για χιλιάδες κτηνοτρόφους λοιπόν οι οποίοι πλήττονται. Ποια είναι η στρατηγική σας και το όρασμά σας ε, βράχει πρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα για να αντιμετωπιστεί αυτή η πανδημία. Πώς μπορούμε να έχουμε μέτρα για να το καταπολεμήσουμε και να έχουμε και μέτρα ε, βιοασφάλειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Καταρχάς θέλω να είμαι απόλυτα σαφής γιατί θεωρώ ότι η υγεία και η ευημερία των ζώων είναι τμήμα της ε, υγείας ε, σε όλα ε, είναι ένα απόσπαστο τμήμα και δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ε, ασήμαντο. Η πανόλη των χείρων είναι μια καταστρεπτική ασθένεια. Δεν αφορά τους ανθρώπους βεβαίως, αλλά αποτελεί απειλή για την ε, πολύτιμη κτηνοτροφία και φυσικά και για το εμπόριο. Είναι παγκόσμια ανησυχία ακόμα. Να σας πω όμως, και αυτό διαφέρει λίγο από τη θέση ε, την οποία δηλώσατε εσείς, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα εύρωστο νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένη πολιτική από αυτό και έχει καταφέρει να περιορίσει την πανόλη των χείρων μόνο σε κάποιες περιοχές. Το παράδειγμα της Τσεχικής Δημοκρατίας, για παράδειγμα, στην οποία εκριζώθηκε η νόσος. Ε, σε άλλες περιοχές, ε, επειδή ακριβώς είναι πολύ κοντά στα σύνορα με άλλες χώρες οι οποίες πλήττονται, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι, να αυξηθεί η βιοασφάλεια στις ε, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η έρευνα, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για την ασθένεια αυτή και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί στο φωτεινό υπόδειγμα ε, για να μην υπάρχει εξάπλωση μιας ασθένειας η οποία μπορεί να επηρεάζει μεν ε, ε, τους χείρους και τους αγριόχειρους αλλά είναι ολέθρια τα αποτελέσματα για όσους ζουν σε αυτές τις περιοχές και φυσικά για τους κτηνοτρόφους της εκμεταλλεύσεις τους. Το γνωρίζω απόλυτα το θέμα και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, ο οποίος ε, στόχο έχει να παρέμβει με συντονισμένο τρόπο όταν υπάρχουν πυρκαγιές και πλημμύρες. Και αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν υποστήριξη ε, και εξοπλισμό και επιμελητία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις κρίσης. Θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο σε περίπτωση επιδημία, σε μεγάλη κλίμακα για ε, κτηνιατρικές νόσους ε, και ζωονόσους γενικότερα. Μπορούμε ε, να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές, για παράδειγμα, με εμβολιασμό σε μεγάλη κλίμακα σε περιοχές που πλήττονται. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κάποιος την εξάπλωση μιας ασθένειας αν εμφανιστεί σε μια περιοχή ή κάπου όπου διαμένουν φυσικά και άνθρωποι. Ευχαριστώ. Υπάρχει παρέμβαση σε περίπτωση κρίσης, ε, όταν υπάρχουν επιδημίες ή ζωνώση, που και μάλιστα έχει υπάρξει και ιδιαίτερα αποτελεσματική. Γιατί στην περίπτωση της Αφρικανικής ε, ε, Πανόλης των Χείρων, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να περιορίσει την εξάπλωση της νόσου σε κάποιο βαθμό. Πρέπει να δρούμε αμέσως όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε το συντομότερο δυνατόν την κατάσταση να πω και κάτι το οποίο δεν έχει προκύψει στη συζήτηση μέχρι τώρα, αλλά μπορεί και να ανακύψει. Ε, είναι ένα πρόβλημα που είχαμε όχι με την ε, υγεία των ζώων, αλλά με την ε, φυτοϊγεία στην Ιταλία, με την ξυλέλεια, στην ελιά. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πλήττει τις ελιές και πολλές άλλες περιοχές, όχι μόνο την Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιήθηκε και έλαβε συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση της ξυλέλεια. Ε, τα κράτη-μέλη βέβαια πρέπει να είναι εξοπλισμένα για να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, ώστε στο μέτρο του δυνατού να δραστηριοποιούμαστε αμέσως και φυσικά να υπάρχει και ένα σύστημα αντιμετώπιση κρίσεων το οποίο θα υπάρχει άμεσα για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατόν. Μακάρι να μπορούσα να σας απαντήσω και να σας πω ότι θα εκριζώσουμε την ε, Αφρικανική Πανόλη των Χείρων στους επόμενους μήνες. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Οι χώρες οι οποίες δεν είναι εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο έχουν πολύ σημαντικότερο πρόβλημα και υπάρχει εξάπλωση και αυτό ίσως ε, σημαίνει ότι και οι χώρες που έχουν σύνορα με αυτές τις χώρες θα έχουν πρόβλημα ακόμα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να μας απασχολεί γιατί αφορά τις ε, κτηνιάτρους, την κατάλληλη κτηνοτροφία και, τις, ε, και το εμπόριο. Ο Ζωάο Φερέρα από την Κούρα. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Αναφερθήκατε στα φυτοφάρμακα και στη διαδικασία έγκρισή του τους γνωμημένους οργανισμούς, την ευαισθητική ασφάλεια, τα φάρμακα. Είναι διάφοροι τομείς όπου εδώ και χρόνια έχουμε στοιχεία ότι οι διάφοροι φορείς της Ένωσης και η Ένωση έχουν υπερβολικά στενές επαφές ε, με τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ορισμένοι φεύγουν από θέσεις υπευθύνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά γίνονται στελέχη αυτών των επιχειρήσεων. Και αυτό επηρεάζει και τη διαδικασία έγκρισης διαφόρων ουσιών. Αυτό μας δημιουργεί πολλές υπόνοιες ε, για το κατά πόσο είναι αυστηρή διαδικασία έγκρισης και κατά πόσο είναι σωστές και διαδικασίες αξιολόγησης της χρήσης μετά. Τι σκέφτεστε για αυτές τις ε, υπερβολικά στενές σχέσεις ε, πιστεύετε ότι μπορείτε να εξακολουθήσετε ε, να πιστεύετε τις ε, αναλύσεις κινδύνου που προκύπτουν από τον ίδιο τον κλάδο. Δεν θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα εμείς ως δημόσιες αρχές να συμμετέχουμε πιο άμεσα στη διαδικασία έγκρισης ουσιών, να έχουμε δηλαδή και τις δικές μας αναγκαίες αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μα κατανοώ πλήρως ότι ορισμένες φορές υπάρχει κάποια δυσπιστία για κάποιες αποφάσεις που λαμβάνουν διάφοροι ευρωπαϊκοί φορείς, όπως ο ε, Οργανισμός Ασφαλεία Φαρμάκων, Ασφαλείας Φαρμάκων. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ελέγχεται και από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά και από το κοινοβούλιο αυτός ο οργανισμός, η ΕΦΣΑ. Και υπάρχουν και πολύ αυστηροί κανόνες για το πώς οι επιστημονικοί φορείς της ΕΦΣΑ, τα μέλη τους δηλαδή, πρέπει να ενημερώνουν τα Μητρώα για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Εγώ εμπιστεύομαι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Χρειαζόμαστε για πολλά πράγματα οι αξιολογήσει να είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα, κάποια προϊόντα, κάποιες ουσίες, αλλά ξέρω ότι έχω την πολιτική ευθύνη για την ΕΦΣΑ και δεν θα είχα καμία αμφιβολία αν θεωρούσα ότι τίθε το θέμα αξιοπιστίας των ε, αξιολογήσεων της ΕΦΣΑ να διερευνήσω εγώ ίδια το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σημειώνω την απάντησή σας. Αλλά θα ήθελα να επεκταθείτε λιγάκι. Δηλαδή, οι απαντήσεις σας ε, δεν είναι ικανοποιητικές για το εξής. Είναι για τη διαδικασία αξιολόγησης, ιδιαίτερα για τα φυτοφάρμακα. Ερώτηση λοιπόν, πώς θα διασφαλίσετε ότι οι αναλύσεις κινδύνου λαμβάνουν υπόψη όλα τα αποτελέσματα, όχι μόνο τα άμεσα αλλά και τα χρόνια. Για τα φυτοφάρμακα πάντα. Συνεχίζω. Πώς θα διασφαλίσουμε να μην μπαίνουν από την πίσω πόρτα ορισμένα φάρμακα που δεν εγκρίνουμε ή φάρμακα που περιέχουν τα τρόφιμά μας λόγω των συμφωνιών ελευθερομπορίου. προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν σας έπεισα για τα φυτοφάρμακα. Γιατί είναι ένα τομέα που είπα ότι θα δεσμευθώ για μείωση των φυτοφαρμάκων και για έγκριση χαμηλού κινδύνου εναλλακτικών ουσιών. Δεν σας έπεισα, προφανώς. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας, είναι τμήμα της Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής από τη φάρμα στο πιάτο. Και είπαμε επίσης ότι θα περιμένουμε για κάποιες αξιολογήσεις που πρόκειται να εκπονήσει η ΕΦΣΑ και θα αποφασίσουμε βάσει τα στοιχεία αυτά. Κάποιος συνάδελφός σας αναφέρθηκε στη σημασία της λήψης επιστημονικών, της λήψης υπόψης επιστημονικών στοιχείων. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλήσαμε για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, τα νέο νοικοτινοειδή, νέες ε, τεχνικές εκτροφής. Όλα αυτά πρέπει να τα εξετάζουμε με βάση τα στοιχεία. Ο Γενικός Νόμος για το Τρόφιμα νομίζω ότι θα αυξήσει τη διαφάνεια, θα αντιμετωπίσουμε ένα από τα αίτια της δυσπιστίας των πολιτών. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Βεβαίω είπα ότι πρέπει να μειωθεί η εξάρτησή μας από τα φυτοφάρμακα και να βρούμε εναλλακτικέ χαμηλού κινδύνου. Αυτό είναι το τμήμα της στρατηγικής μία υγεία. Τμήμα της στρατηγικής από το κτήμα στο πιάτο. Τμήμα της στρατηγικής της πράσινης συμφωνίας. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε από κοινού την ε, υγεία των ατόμων, των ζώων και του περιβάλλοντος και των φυτών. Αλεξάνδρα Μορέτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ υποψήφια, μια ισορροπημένη διατροφή είναι ουσιαστική για την πρόληψη κάποιων ασθενειών, μεταξύ των οποίων κάποιοι όγκοι, καρδιαγγειακές ασθένειες και ο διαβήτης. Και να προλάβει την ε, παχυσαρκία των παιδιών όλο και πιο εμφανή στην Ευρώπη. Συμφωνείτε ότι για να μπορέσουν οι καταναλωτές να κάνουν υγιεινές επιλογές είναι σημαντικό να τους ενημερώνουμε με διαφανή τρόπο, να βασιζόμαστε σε επιστημονικά στοιχεία και να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε προγράμματα εκπαιδευτικά για την διατροφική ασφάλεια. Πώς θα φρενάρετε διάφορα συστήματα επισήμασης των τροφίμων που χρησιμοποιούνται θελοντικά σε πολλά κράτη-μέλη. Θεωρείτε ότι ένας τρόπος επισήμασης ε, στη βασική συσκευασία ε, είναι, θα μπορούσε να είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα. Θα παρουσιάσετε μια πρόταση ούτως ώστε ο καταναλωτής να έχει πληροφορίες για την περιβαλλοντική επίπτωση των τροφίμων και σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται παραδοσιακοί γάματα φόμικρον σε ζωοτροφές. Επίσης, οι ισχυρισμοί για την υγεία. Μερικές φορές ισχύζονται ότι κάποια τρόφιμα έχουν θετικές επιπτώσεις τελείως φανταστικές στην ανθρώπινη υγεία. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Είναι παράδοξη η εποχή μας. Δεν είναι. Μιλάμε για την παχυσαρκία και τώρα παράλληλα αντιμετωπίζουμε ότι έχουμε και πρόβλημα με τη σπατάλη των τροφίμων. 20% των τροφίμων μας τα πετάμε. Ένας από τους τέσσερις όμως Ευρωπαίους δεν μπορεί να έχει ποιοτικό γεύμα με στη μέρα του. Πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Και θα ήθελα να μπορέσω να κάνω κάτι, ούτω ώστε να έχουμε αυτό το πενταετέ ε, σχέδιο δράση για να αντιμετωπίσουμε τη σπατάλη των τροφίμων, γιατί είναι πολύ σημαντικό τμήμα μιας προσπάθειας για βιώσιμα τρόφιμα. Αναφέρατε την ε, επισήμαση για τη θρεπτική αξία. Είναι υποχρεωτική σε συσκευασμένες τροφές. Το θέλουν οι καταναλωτές. Θέλουν τέτοια προφίλ. Όταν παίρνουν κάτι από το ράφι, ψάχνουμε και διαβάζουμε να δούμε αν το προϊόν αυτό έχει τα συστατικά που θέλουμε για να το αγοράσουμε. Ο πρόσφατος καονισμός για τους διατροφικούς ισχυρισμούς λέει ότι μερικές φορές αυτά που διαβάζουμε στην ετικέτα δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Έχουν, ας πούμε, πάρα πολύ ζάχαρη ή αλάτι. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. το διατροφικό προφίλ είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Υπάρχει μια έκθεση για την, το προστινό μέρος της συσκευασία που θα βγει φέτος. Περιμένω να δω τα αποτελέσματα για να προχωρήσω. Και θα ήθελα να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, αν αυτό θα είναι το Nutri-Score ή όχι, δεν ξέρω. Πάντως αυτό είναι ένα θέμα που θα με απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Σταθήκατε και περιγράψατε το πρόβλημα. Πώς θα αποτρέψετε τις τρευλώσεις στην εσωτερική αγορά και θα εγγυηθείτε ότι οι καταναλωτές δεν θα παραπλανώνται από πολύ απλουστευτικές ε, περιγραφές που τελικά οδηγούν και σε διακριτικές ε, μεταχειρήσεις ε, εις βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων αριστείας. Τι σκέφτεσαι συγκεκριμένα για να εφαρμόσετε ένα ενιαίο σύστημα για την επισήμανση των τροφίμων και κυρίως για την προστινή ε, συσκευασία. Έχουμε θαυμάσια επίπεδα ελέγχων στην ενιαία αγορά για να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ούτως ώστε να ξέρουμε, και είναι πολύ σημαντικό για να ξέρουμε και τι μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα ήδη ότι θα περιμένω τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το προστινόμενο της συσκευασία για να αποφασίσω αν θα υποβάλω πρόταση. Αλλά όπως σας είπα, με απασχολεί το θέμα των διατροφικών ισχυρισμών και υπάρχει και ο σχετικό κανονισμό. Κάτι που δεν είπα και θέλω να το πω. Πολλοί καταναλωτές και πολίτες ζητούν να υπάρχει επισήμανση της προέλευσης. Σε 7 κρατημέλη έχει προκύψει αυτό. Και έχουν προχωρήσει από μόνα τους. Και έχουν διαφορετική επισήμανση τώρα για την προέλευση των τροφίμων. Αυτά τα 7 κρατη αξιολογούν τη στάση τους, τα μέτρα τους. Θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν θα πρέπει να επανεθνικοποιήσουμε τα τρόφιμα στην ενιαία αγορά θα πρέπει να βρούμε κοινού τρόπου, ούτως ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφορία όταν αγοράζουν τρόφιμα. Ή καταναλώνουν τρόφιμα. Αυτό το είναι σε φάση αξιολόγησης, θα δω όλες τις σχετικές πληροφορίες και θα υποβάλω ενδεχομένω πρόταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Άουκεν από τους Πρασίνους. Εδώ είμαι. Αξιότιμη υποψήφια επίτροπε. Ένα από τα θέματα τα οποία επιβαρύνει περισσότερο τον εθνικό προπολογισμό για την υγεία είναι οι καταχρηστικά υψηλές τιμές στα φάρμακα, ενώ τα κράτη-μέλη είναι σε ασθενή διαπραγματευτική θέση λόγω της έλλειψης διαφάνειας στη δημολόγηση. Το 2017 ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση για πρόσβαση σε φάρμακα και ζητούν διαφάνεια στη δημολόγηση των φαρμάκων, κυρίω ε, όσον αφορά τι διαπάνε για την έρευνα και την ανάπτυξη, πώ από αυτά ε, χρηματοδοτούνται από το δημόσιο προπολογισμό, ποιο τμήμα είναι marketing και εμπορία και ποιο είναι και κέρδος. Ε, δυστυχώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, τηρήσει καμία από αυτές τις απαιτήσει για τη διαφάνεια. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και άλλα κράτη-μέλη υποστήριξαν ε, ένα ψήφισμα ε, για τη διαφάνεια στη τιμολόγηση των φαρμάκων που θα υποχρεώσει τις φαρμακευτικές εταιρείε να δώσουν στοιχεία για τα όσα σας ανέφερα. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ καλό ψήφισμα. Ωστόσο, το ψήφισμα... Ε, μειώθηκε στην βαρύτητά του πολύ ουσιαστικά και κυρίως και στη χώρα μου στη Δανία ε, και η ερώτησή μου είναι εξή. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι στις διαπραγματεύσεις για την τιμολόγηση των φαρμάκων στα κράτη-μέλη θα υπάρχει δικαιοσύνη και διαφάνεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, να σταθούμε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην πράξη. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο έχει αντίκτυπο στη ζωή των ε, πολιτών και των ασθενών ε, πιο συγκεκριμένα, γιατί υπάρχουν ε, ελλείψεις φαρμάκων και φάρμακα τα οποία δεν είναι προσιτά. Θα συνεργαστώ στενά λοιπόν με τον κλάδο αλλά και με τα κράτη-μέλη, γιατί πρέπει να ε, δούμε και τους μηχανισμούς τιμολέγησης των κρατών μελών και πώς αποζημιώνονται τα φάρμακα, γιατί και αυτό είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει νομική υποχρέωση ο φαρμακευτικός κλάδος ε, να δίνει πρόσβαση σε στοιχεία ε, για την ε, παρασκευή φαρμάκων και πρέπει να εξετάσουμε μια νέα στρατηγική που θα αντιμετωπίσει και τις ελλείψεις των φαρμάκων αλλά και την τιμολόγηση. Και θα συνεργαστώ πολύ στενά με τα κράτη-μέλη για να το εξετάσουμε το θέμα αυτό, διότι το πρόβλημα που υπάρχει με την τιμολόγηση και την αποζημίωση στην ουσία επηρεάζει και την εφαρμογή της οδηγίας για τους διασυνοριακούς ελέγχους και το πώς υπάρχει πρόσβαση ασθενών σε αυτή ε, τον έλεγχο. Θα το εξετάσω λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικά με τα κράτη-μέλη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Επίσης γνωρίζω ότι τα κράτη-μέλη έχουν συστήσει μια task force με τον EMA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αν δεν κάνω λάθος, ε, είμαστε εν αναμονή της έκθεσης η οποία λογικά θα μας δώσει και πολύτιμες πληροφορίες. Με βάση αυτό θα αποφασίσω και τι μέλη γενέστε. Συμφωνώ όμω μαζί σας ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και στην επιστολή για την αποστολή μου τα προσιτά φάρμακα αναφέρονται ρητός. Σίγουρα λοιπόν θα είναι υψηλά στις προτεραιότητές μου. Ε, το θέμα όμως έγινε πιο περίπλοκο από την ερώτηση. Η ερώτησή μου ήταν πάρα πολύ απλή. Και αν ε, το δείτε και μπορείτε να το κάνετε, γιατί ξέρω ότι ο Πόη ε, διαρρέει πράγματα, γιατί ήταν, ε, διέρευσαν κάποια πράγματα για τα όσα γίνονταν στο ΠΟΕ, γιατί ήταν εμπιστευτικέ οι πληροφορίε. Αλλά το θέμα είναι ε, τι γίνεται. Στι χώρε ε, τελικά υποκύπτουν στι μεγάλε βιομηχανίε. Αυτό έγινε στη Δανία και στη Γερμανία και σε άλλε χώρε. Θα ήταν πολύ χρήσιμο όμω για τα κράτη-μέλη που βλέπουν τι τιμέ να εκτοξεύονται κάθε χρόνο. Και πραγματικά αυτό καταστρέφει νοσοκομεία, και μειώνει φυσικά και ε, τις διαδικασίες και υπάρχει μια μακριά διαδικασία, αλλά να δούμε την πραγματικότητα. Απλές ερωτήσεις. Ε, εξασφαλίστε ότι θα υπάρχει διαφάνεια στην τιμολέωγηση. Τελεία και παύλα. Λυπάμαι που περιέπλεξα την ερώτησή σας. Ε, ίσως δεν έχω εύκολη απάντηση. Αλλά εγώ υποστηρίζω τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Ε, πρέπει να το εξετάσω πιο προσεκτικά. Υπάρχει περίπτωση να μην είμαι τώρα ε, σε θέση να σας απαντήσω γιατί δεν διαθέτω όλες τις πληροφορίες και να επανέλθω. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής λοιπόν επ' αυτού. Ευχαριστώ. Νικολάη Στεφανούτα από το Renew Europe. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, θα συνεχίσω με τις ερωτήσεις κυρίας Κοπάτς και Άουκεν και θα μιλήσω για την έλλειψη Ίσως επαναλάβω τα ίδια και τα ίδια, αλλά θέλω να ξαναβάλω κάποια επιχειρήματα. Από το καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε μια τεράστια κρίση στην Ιταλία, για... στην Πολωνία, στην Ιταλία φάρμακα καρκίνου, νευρολογικά φάρμακα στην Πολωνία, γενικά φάρμακα στο Βέλγιο δεν υπάρχουν, επίσης στη Ρουμανία ε, οι μουνογλομπίνες έλειπαν και ζητήσαμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Προστασίας, ο οποίος είναι απόδειξη ότι πρέπει να είσαι πολύ εφάνταστος, ούτω ώστε να είναι αποτελεσματική για τους πολίτες η πολιτική υγείας. Και φτάνω στην ερώτησή μου. Κάτι που δεν αναφέρθηκε σήμερα ήταν το Brexit, το οποίο έχει σημασία όταν μιλάμε για τη διαθεσιμότητα φαρμάκων στην αγορά. Το ερώτημά μου ή τα ερωτήματά μου είναι, θα μας πείτε αν δεσμεύεστε για να αναπτυχθεί ένας κατάλογος ευρωπαϊκών ουσιαστικών ή βασικών φαρμάκων, θα προτείνεται νομοθεσία για την έγκαιρη προειδοποίηση για τις ελλείψεις των φαρμάκων. Κάπως το αναφέρατε νομίζω, αλλά τι θα κάνετε με τα επίγοντα και επειδή αναφέρατε την αγορά ως λύση σε πολλές από τις απαντήσεις που δώσατε πριν. Θέλουμε όλοι να μάθουμε αν θα γίνουν θα είσαστε επίτροπο που θα κάνει παρεμβάσει, θα είσαστε εφάνταστο ε, επίτροπο Ή θα είστε ένα κλασικό επίτροπο. Φαντάζομαι ότι η τρίτη εναλλακτική δεν είναι η σωστή εναλλακτική. Καταρχά, πρέπει να γίνω πρώτα επίτροπο για να κάνω οτιδήποτε. Και μετά σα αφήνω να κρίνετε τι είδου επίτροπο είμαι. Γιατί μπορεί εγώ να νομίζω ότι θα είμαι ο Α τύπο ή ο Β τύπο και εσεί να έχετε άλλη άποψη. Α κρίνετε εσεί λοιπόν τι είδους επίτροπος θα είμαι αν γίνω. Αναφέρα, ανέφερα την Task Force στην πολύ περίπλοκη απάντηση που έδωσα πριν. Η Task Force δημιουργήθηκε από τα κράτη-μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ούτω ώστε να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τις ελλείψεις στα φάρμακα. Και ανέφερα ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και ότι πρέπει να βρούμε ένα σύστημα για την έγκαιρη προειδοποίηση για τις ελλείψεις που υπάρχουν στα φάρμακα. Ξέρω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αποφύγουμε το θέμα του Brexit. Είναι κάτι που απασχολεί ε, πολλούς, πολλά κρατημέλη γιατί μπορεί να σχετίζεται με το κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα λόγω του Brexit. Υπάρχουν ανησυχίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και τα κρατημέλη μελη ζήτησαν οι εταιρείε να υπαγρυπνούν γιατί πρέπει να γίνονται έλεγχοι κεντρικά των φαρμάκων. Υπάρχουν όμως και κάποια φάρμακα που τα εγκρίνουν οι εθνικές αρχές. Εκεί υπάρχουν προβλήματα. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμα αυτά τα φάρμακα μετά το Brexit. Για δύο χώρες υπάρχει το πρόβλημα. Τη δική μου χώρα που ξέρω καλύτερα και τη Μάλτα. Αυτό που θα ήθελα να συμβεί είναι μια επικύρωση της συμφωνίας ε, αποχώρησης, ούτως ώστε να έχουμε ελάχιστε διαταραχές σε όλους τους τομείς, καθώς και σε αυτόν της πρόσβασης στα φάρμακα. Μετά από αυτό που είπατε για την Task Force, δεν θα ήταν καλύτερο αντί να περάσουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να υπάρχει μία ε, ένας οργανισμός ευρωπαϊκός ε, που θα αντιμετωπίζει τη ελλείψεις των βασικών φαρμάκων μέσω συντονισμού των προσπαθειών σε κάποιες πλατφόρμες. Ο συνάδελφος μου είπε βέβαια ότι δεν θα πρέπει να σταθώ στην τυπική ουσία του Brexit. Όχι, δεν το ανέφερα με τυπικό τρόπο, είναι μια ανησυχία που έχω. Ίσως αυτό που προτείνεται είναι ένα καλύτερο τρόπος να προχωρήσουμε. Αλλά είπα, και μπορεί να σας φανεί ότι επαναλαμβάνομαι, ότι πρέπει να έχουμε πληροφορίες πριν λαμβάνουμε αποφάσεις. Και η Task Force δημιουργήθηκε για να δώσει αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες για τις ελλείψεις. Θέλω να αξιολογήσω τα αποτελέσματα των προσπαθειών της Task Force και μετά θα είμαι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις και θα συμπεριλάβω όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς γιατί πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα που επηρεάζει τους Ευρωπαίους ασθενείς και που ονομάζεται έλλειψη φαρμάκων. Ε, ο τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σπαντικός, ο Πέτρα Λίζα. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, το σημαντικό θέμα που ήθελα να θίξω έχει διαπαντηθεί και με ικανοποιεί η απάντησή σα. Κοιτάξτε, είναι σαν τη μέρα με τη νύχτα με την ακρόαση που κάναμε σήμερα το απόγευμα. Είμαι λοιπόν ικανοποιημένο αλλά έχω και άλλε ερωτήσει. Συγκεκριμένη ερώτηση για την αντίσταση σε αντιβιωτικά. Δύο προκλήσει νομίζω αντιμετωπίζεται. Πρώτον, η εφαρμογή τη νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Το Κοινοβούλιο πίεσε πολύ ότι τα αντιβιωτικά τελευταίας καταφυγής ή θα πρέπει να απαγορευτούν ή θα πρέπει η χρήση τους να περιοριστεί πάρα πολύ. Είστε διατεθειμένοι να τα απαγορεύσετε στο μέτρο του δυνατού είναι η πρώτη ερώτησή μου, όπως ήθελε το Κοινοβούλιο. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως νέα αντιβιωτικά. Είπατε θέλετε να ενθαρρύνετε μαζί με τις φαρμακοβιομηχανίες την ανάπτυξή τους. Αλλά υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, όπως για παράδειγμα για τα παιδιατρικά φάρμακα, δηλαδή και κυρώσεις και κίνητρα. Να βοηθήσουμε, να δώσουμε κίνητρα λοιπόν στις φαρμακοβιομηχανίες για να ε, βρουν νέα φάρμακα, αλλά να έχουμε και κυρώσεις για να τις ε, ενθαρρύνουμε ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Λίζε. Ναι, με η τελευταία ερώτηση, αλλά νομίζω ότι είναι από τις πιο μεγάλες προκλήσεις. Κοιτάξτε. Πρώτον, Έχουμε τον κανονισμό του 2018, νέο κανονισμό, για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο στοιχείο της αντιμετώπισης της ε, αντίστασης στα αντιβιωτικά στα ζώα. Επίσης, έχουμε μια οδηγία που λέει ότι γενικά πρέπει να απαγορεύονται για την ε, κτηνοτροφία και ορισμένα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ασθενείς ανθρώπους. Τώρα πώς εφαρμόζεται. Έχουμε ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων και επισκέψεων στα κράτη-μέλη. Να δούμε πώς θα πάει. Αναφέρθηκα στον κλάδο και στην καινοτομία. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ακριβώς να ηγείται μέσω βελτίστων πρακτικών για να έχουμε νέα τέτοια αντιβιωτικά. Επίσης, θα ήθελα να εκδοθεί η αξιολόγηση για τα ορφανά και παιδιατρικά φάρμακα για να δούμε πού τα πήγαμε καλά, πού δεν τα πήγαμε καλά πριν προτείνω κάτι παρόμοιο ή κάτι διαφορετικό. Το θέμα δεν είναι πάντα να υπάρξει νέα νομοθεσία είναι πολλές φορές θέμα εφαρμογής της υπάρχουσας. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τα δύο αυτά θέματα. Οπότε ο κανονισμός για τα παιδιατρικά και ορφανά όντως έσωσε ζωές και άλλαξε τις ζωές πολλών παιδιών με σπάνιες ασθένειες. Τώρα αξιολογείται η χρήση του. Θα δούμε τη λέει αξιολόγηση και μετά θα δούμε εάν πρόκειται να προτείνουμε περαιτέρω νομοθεσία. Πολλά κράτη-μέλη συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε νέα αντιβιωτικά και καινοτομία. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να παίξει ρόλο η Ευρώπη σε αυτό. Συμφωνείτε ότι επειδή η αγορά σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ίσως επαρκώς ελκυστική για τις φαρμακοβιομηχανίες, χρειαζόμαστε, συμφωνείτε λοιπόν, ότι χρειαζόμαστε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αντιδράσεις των κρατών μελών σε αυτό. Μα ήδη είπα ότι θέλω να μιλήσω για το μέλλον, αλλά τώρα θέλω να μιλήσω και για το παρελθόν, γιατί η Επιτροπή το 2017 πρότεινε το δεύτερο πρόγραμμα δράσης για την ε, καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντίστασης. Τώρα, με το θεματολόγιο για τη μία υγεία που είναι μέσα στην επιστολή μου, με συγχωρείτε που το το έχω πει επανειλημμένα, είναι πολύ σημαντικό. Και καταλαβαίνω ότι η πρόκληση είναι για μένα, επειδή η επιστολή καθηκόντων αναφέρει την αντίσταση στα αντιβιωτικά, αναφέρει τους διαταράκτες, αναφέρει το πρόγραμμα για τον καρκίνο, αναφέρει το πρόγραμμα από το κτήμα στο πιάτο. Πρέπει λοιπόν με υπεύθυνο τρόπο να τα προωθήσουμε όλα αυτά. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, αλλά ναι. Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπαθία, διότι το πρόβλημα αντίσταση στα, μικρο, στα αντιβιωτικά είναι παγκόσμιο. Χρειάζεται κοινή δράση. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί αυτής της προσπαθίας. Ωραία, οπότε τα δικά σας πορίσματα. Έχετε πέντε λεπτά. Αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να τα εξαντλήσετε. Να θεωρήσω ότι αυτό σημαίνει ότι καλύτερα να μην μιλάτε πέντε λεπτά, αλλά Καταρχάς δεν θα μιλήσω για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για το χρόνο και τις ερωτήσεις σας. Τις ε, περασμένες εβδομάδες ε, άκουσα πολλούς να λένε ότι αυτή η ακρόαση θα είναι τρομακτική εμπειρία και σας διαβεβαιώ ότι δεν ήταν ε, και περίπατος. Αλλά ε, υπήρξε πρόκληση και πρέπει να πω ότι απόλαυσα το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση πολιτικής για αυτό το οποίο πραγματικά ελπίζω ότι θα είναι το χαρτοφυλάκιό μου. Μίλησα με ειλικρίνεια και ε, γνωρίζετε ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το χαρτοφυλόκιο. Δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου να βρίσκομαι εδώ εάν δεν πίστευα σε κάτι τέτοιο και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα μαζί. Και αυτό γιατί το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αφορά την καθημερινή ζωή των πολιτών, αφορά την υγεία τους, αφορά την ε, ζωή τους και αφορά τα τρόφιμά τους. Και όταν ε, αναφέρομαι στο χωράφι, στο πιάτο ή μία υγεία, μία προσέγγιση για την υγεία, αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά λόγια για μένα, είναι η ουσία, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Άκουσα τις ανησυχίες σας, ε, τα άκουσα προσεκτικά. Ενδοκρινικοί διαταράκτες, ε, μικρόβα και εντοχή, αναπαραγωγικές τεχνικές και τα λαμβάνω πλήρως υπόψη, είναι κάποια εξ αυτών που ακούσαμε. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή αυτή τη στιγμή και οι πολλοί πολίτες περιμένουν από εμά, όλους εμάς, να είμαστε στην πρώτη γραμμή και να κάνουμε αλλαγές και πρέπει να προφυλάξουμε τα επιτεύγματά μας και τα οικοσυστήματά μας για τις μελλοντικέ γενναίες δεν βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να τρανίσουμε. Το οφείλουμε στους πολίτες και το οφείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι τεράστια τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να υπάρξουν οι απαραίτητες ε, λύσεις ε, σε στενή συνεργασία μαζί σας, αλλά να παραδεχτώ ότι έχω και πάρα πολλά πράγματα να μάθω ακόμα. Σας διαβεβαιώ όμως ότι θα ξεκινήσω τρέχοντας εάν ε, επιβεβαιωθώ σε και πάντα θα εργαστώ με διαφάνεια, με επικοδομητικό τρόπο ε, στη συνεργασία μου μαζί σας, διότι ε, στο κάτω-κάτω της γραφής είμαστε υπόλογοι προς εσάς. Με αυτό λοιπόν θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου και να πω ε, κάτι, μια σύντομη δήλωση. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορούμε πλέον να μιλούμε για τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, την ε, υγεία των ζώων και τη φυτοϊγεία και να τα εξετάζουμε μεμονωμένα. Ε, μπορεί να φαίνονται ότι είναι ξεχωριστά νησιά, αλλά στην πραγματικότητα συνδέονται άρρηκτα και οι πολίτες απαιτούν να τους δώσουμε αποτελέσματα. Υπάρχει ένας κοινός στόχος ε, μία υγεία για όλους. Πρέπει να συνεργαστούμε προ όφελο των πολιτών μας. Πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει η κοινωνία των πολιτών και οι πολίτες. Πρέπει να εξετάσουμε περισσότερες επιστημονικές ενδείξεις και θα μοιραστώ κάτι το οποίο πιστεύω ακράδαντα μαζί σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει μάχη για περισσότερα. Να σα ευχαριστήσω και πάλι για το χρόνο σα. Περίπου 3,5 λεπτά μίλησα κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε στενά.